Äh, Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Δεν αρχίζουμε και εντελώς ε, στην ώρα μας, αλλά σχεδόν. Τι έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Λάβατε την πρόσκληση έγκαιρα όλοι. Υπάρχουν παρατηρήσεις στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Και Κατά δεύτερο λόγο πάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Οι συνάδελφοι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές για το COP17 και το σχετικό ψήφισμα κατέληξαν κάπου και έχει υπογραφεί το κείμενο και στάλει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Οπότε είναι και αυτό εντάξει. συγγνώμη. Εδώ η γραμματεία μου επισημαίνει ότι επισήμως και τυπικός, για να μην γίνει λάθος, στα διάφορα, στο τέλος της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να λάβουμε απόφαση ότι αυτό που επεξεργάστηκαν οι εισηγητής και η ε, Σκιώδης ε, αποφασίστηκε επίσημα. Υπάρχει και στην ημερήσια διάταξη και ξέχασα να σας το πω, έτσι όμως θα γίνει. Τώρα, τα πρακτικά. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Τα έχετε μάθει όλοι απ' έξω. Ωραία, προχωρούμε λοιπόν και πάμε στο τέταρτο σημείο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, τον ΕΝΙΖΑ. Ο καθηγητής Τσίτσεστερ είναι ο εισηγητής και του δίνω αμέσως το λόγο. Giles. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, συζητάμε το Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Θυμίζω ότι δημιουργήθηκε ο οργανισμός αυτός κάποιο ε, κάποια χρόνια πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 90, τα ανήσυχα χρόνια, όπως τα λέμε και επεκτάθηκε η εντολή κατά την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου το 2008 και φέτος πάλι ε, δώσαμε παράταση στην εντολή του οργανισμού για να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να εξετάσουμε την πιο ε, ουσιαστική πρόταση από την Κομισιόν για νέο ε, σχεδιασμό της εντολής του οργανισμού. Και Υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα καταρχήν που πρέπει να θέσουμε και το θεμελιώδες είναι ο οργανισμός πρέπει να συνεχιστεί, έχει σκοπό και ένα δεύτερο ερώτημα ανάλογα με την απάντηση στο πρώτο είναι πώς ο φορέας αυτός θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Αναθέσαμε μια μελέτη την οποία ελάβαμε τον Ιούλιο και διοργανώσαμε και στην Επιτροπή μας μια ακρόαση όπου ακούσαμε πολλά στοιχεία για το ρόλο, τη φύση, τις αρμοδιότητες του οργανισμού και τι ε, αλλαγές θα έπρεπε ενδεχομένω να γίνουν. Μετά από όλα αυτά καταλήξαμε ότι ναι, χρειάζεται αυτός ο οργανισμός, πρέπει να συνεχιστεί, αλλά όχι με την ίδια μορφή όπως υπάρχει σήμερα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή στη μορφή του, στο σχήμα του, διότι υπάρχουν σημαντικοί στόχοι, σημαντικά επιχειρησιακά θέματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας που δεν είναι ικανοποιητικά. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε την εντολή ώστε να προβλέψουμε καλύτερη διοικητική δομή, καλύτερη διαχείριση, να θεσπίσουμε σαφέστερες προδιαγραφές για τους γενικούς και ειδικούς στόχους και τα καθήκοντα του οργανισμού και να κάνουμε αλλαγές για να βελτιώσουμε, όπως είπα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, που δείχνει τη δυσκολία του οργανισμού. Το προσωπικό είναι περίπου 60-70 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εκεί απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις. Αυτοί που κάνουν την καθαυτό δουλειά με τους υπολογιστές, ασφάλεια διαδικτύου και υψηλής τεχνολογίας πράγματα είναι μια ντουζίνα. Λίγοι, λίγοι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να κάνουν πολλά ταξίδια για να συναντούν τους ομολόγους τους στα κράτη-μέλη, να δημιουργούν δίκτυα, ε, αφού είναι οργανισμός δικτύων, να δημιουργούν δίκτυα επαφών με ομολόγους, γιατί είναι υψηλή ειδίκευση άνθρωποι που πρέπει να συνομιλούν μεταξύ τους. Και ζούμε βέβαια στην εποχή της πληροφορίας Έχουμε το διαδίκτυο ευρεία ζώνη, ε, βίντεο, βίντεο κλπ. Πάντως ε, η συνάντηση τέτα τέτ ε, είναι πολύ καλή. Για φανταστείτε να κάναμε, σε αυτή τη, να, να, να κάναμε τη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και να καθόμαστε στο σπίτι μας και να μιλούσαμε με το Skype. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και τόσο αποτελεσματικό αυτό. Δεν αντικαθίσταται εύκολα η άμεση επαφή. Χρειάζονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί πολλά ταξίδια να κάνουν. Και τώρα, λόγω της έδρας του οργανισμού, αυτό σημαίνει πάρα πολλά ταξίδια. Αυτό το σημείο αναδείχτηκε και στην ε, έκθεση που αναθέσαμε την ε, έρευνα αυτή δηλαδή ε, παρουσιάστηκε ως πρόβλημα ο χρόνος που απαιτείται για τις συναντήσεις. Με βάση αυτή την παραδοχή λοιπόν ε, της ανάγκης για τη συνέχιση του οργανισμού είδαμε τη διοικητική δομή του, καθήκοντα και στόχους και το αποτέλεσμα από τις 120 τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο έκθεσης και που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα εκτελεστικό συμβούλιο ως ενδιάμεσο μεταξύ του διοικητικού και του γενικού διευθυντή και θα πρέπει να καθορίσουμε το ρόλο του οργανισμού, ο οποίος οργανισμός ε, έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει στο ρόλο του, γιατί από τη μία πλευρά θα πρέπει να συλλέγει πληροφορίες ε, για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, όλα τα θέματα σε μια εποχή και σε ένα χρόνο όπου η κυβερνοασφάλεια ε, αποκτά μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα και πρέπει να το κάνει και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τις ε, αρμοδιότητες των εθνικών οργανισμών, των κρατών μελών που δρούν σε αυτόν τον τομέα. που δεν θέλουν ε, επιχειρησιακό οργανισμό. Αυτός ο οργανισμός όμως παίζει ρόλο συντονιστικό. Παίζει το σύνδεσμο μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και των ε, ομάδων, ερευνητικών ομάδων απόκρισης. Έχουν σύνδεσμο, ε, παίζουν το ρόλο συνδέσμου σε πολλά κράτη-μέλη και μοιράζουν, αν θέλετε, τις βέλτιστες πρακτικές, κυρίως στα μικρότερα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, ε, παίζει το ρόλο συνδέσμου ε, προς τρίτες χώρες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Είναι άλλωστε η κυβερνοασφάλεια ένα παγκόσμιο πεδίο δραστηριοτήτων και εκεί παίζει ο οργανισμός αυτό σημαντικό ρόλο. Κατά συνέπεια, χρειάζονται κάποιες αλλαγές στη σημερινή κατάσταση και το πιο αμφιλεγόμενο θέμα σε αυτές τις αλλαγές είναι η έδρα. Διότι το Ηράκλειο Κρήτης είναι πολύ όμορφο, έχω πάει και έμεινα εκεί Μάλιστα ε, μου πήρε πολύ χρόνο να πάω εκεί και μου πήρε πολύ χρόνο να ξαναγυρίσω. Και έτσι πρακτικά το είδα. Και μάλιστα αυτό έγινε το καλοκαίρι που οι πτήσει είναι πιο συχνέ και πυκνές. Η δυσκολία τη έδρα του οργανισμού υπάρχει. Επειδή είναι σε αυτή την ε, τοποθεσία, σε αυτή τη θέση στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι συμβολικά μιλάμε για την θέσπιση ή σύσταση ενός νέου οργανισμού και γι' αυτό θα πρέπει να του δώσουμε και ένα νέο όνομα. Υπάρχει λοιπόν και σχετική τροπολογία στο σχέδιο έκθεσης που λέει να, να ονομαστεί ουνίσα, όχι ενίσα. Γιατί κάποιοι μιλούν για Ένωση Union αντί για Europe. Αντικαθιστούμε το Europe από το, με το Union. Και έχω καταθέσει και άλλη μία τροπολογία που δίνω το ακρονίμιο New NISA που ακούγεται σαν αυτό που προτείνω, μια, ε, ένα νέο οργανισμό για την ασφάλεια δικτύων και πληροφορών, αλλά το νιου ε, σε αυτή την περίπτωση σημαίνει NEU, New European Union κλπ. κλπ. Ε, το βασικό στην τροπολογία είναι ότι η έδρα πρέπει να είναι στις Βρυξέλλες, να είναι εκεί η έδρα. Κατανοώ ότι η πρόταση αυτή θα με κάνει πολύ ε, αντιδημοφιλή στην Ελλάδα. Αλλά η ώμη μου είναι αρκετά φαρδής Άλλωστε η Ελλάδα έχει πολλά άλλα προβλήματα να την απασχολούν αυτή τη στιγμή, αλλά οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο τωρινός διακανονισμός σε σχέση με την έδρα του οργανισμού δεν εξυπηρετεί. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ προτείνω την πιο ριζοσπαστική αλλαγή. Άλλοι μπορεί να καταθέσουν λιγότερο ριζοσπαστικές λύσεις, ενδιάμεσες, χρυσές τομές. Πάντως πρέπει να αλλάξει για να γίνει αποτελεσματικότερος ο οργανισμός. Δεν μπορεί οι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι να ε, ταξιδεύουν τόσο πολύ και να μην έχουν χρόνο να κάθονται μπροστά στον υπολογιστή τους ή ακόμα πιο σημαντικό να συνομιλούν με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη και να είναι όλο στα αεροδρόμια. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ελπίζω οι συνάδελφοι όταν μελετήσουν την, το σχέδιο έκθεσης και δουν τις τροπολογίες και δουν τι εννοούμε σε ό,τι αφορά ορισμό ε, στόχων, σύνθεση της ομάδας των εμπλεκομένων, των συμμετεχόντων, το νέο εκτελεστικό συμβούλιο, σημεία, όχι, τη δύναμη και το ρόλο του Γενικού Διευθυντή και σύμφωνα με τις πρακτικές που ακολουθούμε και σε σχέση με άλλους οργανισμούς θα επεκτείνουμε τις ευκαιρίες του οργανισμού και του Γενικού Διευθυντή ειδικότερα να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να μας ε, παρουσιάζουν εκθέσεις, να συζητούν μαζί μας και να μας ε, χρησιμοποιούν, αν θέλετε, ως ε, λιδία λίθο για να κρίνουν τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Αυτό λοιπόν θα προκαλέσει, ελπίζω, Σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσει. Ελπίζω να είναι θετικέ οι συζητήσει για το ρόλο και τη λειτουργία του οργανισμού. Αν δεν μπορούμε να ε, κάνουμε κάτι για την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την έδρα και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τότε πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο θεμελιώδες ερώτημα. Θα έλεγα στους φίλους της ελληνικές αρχές ότι αν ε, δεν θέλετε αλλαγή, η μη αλλαγή σημαίνει ότι θα καταλήξει το Σεπτέμβριο του 2013 ο οργανισμός και επειδή έχει ρόλο να παίξει θα προτιμούσα να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη, θα φροντίσω να δοθεί χρόνος για όλα τα θέματα 10 το πρέπει να έχουμε τελειώσει με το ζήτημα αυτό. Λάβετε το υπόψη σας. Κρίστιαν ε, Έντερ, πρώτος ε, ομιλητής ο Σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, χτες ε, συμίλησα και με άλλους συναδέλφους και οι συνάδελφοι Τικάου ήταν και άλλοι συνάδελφοι και μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ κάναμε ένα μεγάλο hearing, μια ακρόαση με θέμα κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένα από τα εντυπωσιακότερα και απλούστερα ίσως αποτελέσματα από αυτό το hearing ήταν ε, ε, όταν ρωτήσαμε έναν πρώην hacker και υπεύθυνο για τον κυβερνοχώρο, ποια είναι τα αποτελεσματικά μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη για την ανάσχεση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Μας είπε λοιπόν ότι το επιχειρησιακό μοντέλο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι το μοντέλο που τι είναι. Είναι low risk, high benefit, χαμηλό ρίσκο, υψηλό όφελος. Αυτό είναι το μοντέλο του. Η χτεσινή εκδήλωση μας έδειξε για ποια τάξη μεγέθους μιλάμε. Πρόκειται για μια κρατική απειλή η ασύμετρη αντιπαράθεση επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Γιατί είδαμε ότι και κράτη-μέλη έπεσαν θύματα τέτοιων επιθέσεων. Ε, οι πρωτόγνωρες διαστάσεις αυτού του εγκλήματος ε, παρουσιάστηκαν στην Κορέα, όπου η χρηματαγορά ε, έγινε αντικείμενο επιθέσεων και, κάποια, και είχε πρόβλημα το χρηματιστήριο στην Κορέα. Οπότε πολλές φορές αξιοποιείται ο πόλεμος στον κυβερνοχώρο για να γίνει ασύμετρη αντιπαράθεση. Και είδαμε τι σημαίνει αυτό για όριμες οικονομίες όπως η Ευρώπη, όπου μέχρι τώρα μόνο εκτιμήσεις κάναμε. 250 δις ευρώ χάνονταν λόγω του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και περίπου το 70% όλων των ε, εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο δεν καταλήγουν σε μηνύσεις. Ένας ανακριτής Γάλλος ε, της Eurojust μας είπε ότι οι εισαγγελίε ε, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα, ούτε το νομικό πλαίσιο επαρκεί, ούτε υπάρχουν μέσα ικανά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αν δούμε τη, λοιπόν τη διάσταση που απόκτησε το πρόβλημα θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή ε, στην Ευρώπη επεξεργαζόμεθα λύσεις αλλά δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Ε, είναι ανεπαρκείς και κατακαιρματισμένες οι δομές που διαθέτουμε και ε, εξαιτίας της διάστασης του προβλήματος σήμερα κανονικά θα έπρεπε ο Ενίζα να κλείσει. Για πολλούς λόγους που έχουν σχέση με τα κράτη-μέλη, παλιά είχαμε πει και εγώ τότε ήμουν ένας από τους σκιώδεις εισηγητές, ε, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια συμβιβαστική λύση μεταξύ κρατών μελών και τα, ε, γιατί τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη δεν ήθελαν τον Ενίζα, ενώ άλλα κράτη-μέλη ήθελαν να έχουν ένα θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο το οποίο θα μπορεί να παράσχει υποστήριξη και βοήθεια ε, για να δημιουργηθούν τέτοιες δομές στα κράτη-μέλη. Οπότε ουσιαστικά αν θέλετε έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και η απάντηση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα είναι μια δύσκολη ευρωπαϊκή συμβιβαστική λύση. Αυτή ήταν η απάντηση που βρήκαμε και αυτό πρέπει να αλλάξει καθοριστικά. Το είδαμε με το, την κατάρρευση του Emission Trading Platform, το ETS, είδαμε ότι ένα πολιτικό μέσο ε, έπεσε ε, θύμα ε, με την απώλεια 40 δις ευρώ. Ε, και αυτό έχει να κάνει με τις ληστείες στις τράπεζες. Επανέρχομαι λοιπόν για να υποστηρίξω την ε, δραστήρια παρέμβαση του κυρίου Τσίτσεστερ χρειαζόμαστε αποτελεσματικό ενίζα Χρειαζόμαστε έναν ενίζα ο οποίος θα είναι πολύ πιο ε, στεναρά ενσωματωμένο στην οριζόντια διάσταση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ικανότητες στη Europol, πρέπει να υπάρχει δικτύωση εδώ με, ε, με τον ενίζα. Θέλουμε δομές με τον ε, GRC. Περίπου 300 άνθρωποι ασχολούνται εκεί με την ασφάλεια του διαδικτύου και τώρα διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς χωρίς ανταλλαγές με τον ΕΝΙΖΑ. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα ε, για την ασφάλεια της έρευνας. Τα επόμενα δύο χρόνια θα δαπανηθούν πολλά ε, ε, χρήματα, χωρίς να είναι ο ΕΝΙΖΑ κομμάτι εδώ, γιατί για χρόνια συζητούσαμε το σχέδιο, την ασφάλεια της πληροφορίας χωρίς τον ΕΝΙΖΑ και μάλιστα τώρα δεν έχουμε καν υποχρέωση της Κομισιόν σε, νομοθετή, σε νομοθετήματα ε, να ερωτά την Ενίζα, τον Ενίζα. Δηλαδή ο Ενίζα δεν ερωτάται σε όλα τα ζητήματα. Οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε πιο αποτελεσματικές δομές. Εγώ υποστηρίζω 100% την πρώτη πρόταση της Κομισιόν για την ε, διεύρυνση επέκταση και όλες οι ομάδες με τις τροπολογίες το υποστηρίζουν και πρέπει παραταξιακά διακομματικά να συμφωνήσουμε ότι είτε ότι χρειαζόμαστε νέο οργανισμό ή τον ενίζα να τον διευρύνουμε, να τον κάνουμε αποτελεσματικότερο, να τον ε, εξοπλίσουμε με προσωπικό γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να Δηλαδή θα είναι γελίο το πώς αντιμετωπίζουμε το, τις σημερινές προκλήσεις στο έγκλημα στον κύβερνο χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδελφούς, τόσο τον κύριο Τσίσεστερ, όπως και τον κύριο Μελέρ, όπως και στην κυρία Ντίλαν Βαλεάν, όπως και στον κύριο Λαμπέρτ, για τη συνεργασία που είχαμε όταν συζητήσαμε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση η ομάδα μας ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών υποστηρίζει να υπάρχει ένας ε, ισχυρός οργανισμός με διαπριμένη εντολή που να συμπεριλαμβάνει και το επιχειρησιακό κομμάτι αλλά και το κομμάτι της εκπόνησης νομοθεσίας και το τμήμα της διεθνούς συνεργασίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να υποστηρίξουμε είναι η επέκταση, παράταση, επέκταση της εντολής, με συγχωρείτε, του οργανισμού. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος χαρακτήρας της εντολής. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ορισμένοι από τους εμπειρογνώμονες ε, σε θέματα ασφαλείας πληροφοριών δεν ε, αισθάνθηκαν ε, ότι επιθυμούσαν να εργαστούν στην ΕΝΙΣΑ ακριβώ γιατί έχει αυτή την περιορισμένη εντολή. Έτσι λοιπόν ένας ε, καλός ε, επαγγελματίας δεν πρόκειται να πάει εκεί να εργαστεί γιατί δεν θα έχει μικροπρόθεσμη σταδιοδρομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αποτελεσματικό οργανισμό με διευρυμένη εντολή, έναν ισχυρό οργανισμό. κατά τα Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στρατηγική πολύ αποτελεσματική για το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να συμμετέχουν ε, πάρα πολλά όργανα ε, και ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και εθνικοί θεσμοί. Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες ε, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού να είναι εμπειρογνώμονε ε, σε θέματα πληροφορική. Γι' αυτό έκανα μία πρόταση τροποποίηση προ αυτή την κατεύθυνση για να περιοριστεί στο 40% το διοικητικό προσωπικό. Μόνο δηλαδή το 40% του προσωπικού είναι διοικητικό και οι υπόλοιποι να είναι εμπειρογνώμονες για να καταπολεμούν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Δεν συμφωνώ με το να αλλάξει το όνομα αυτού του οργανισμού όταν μιλάμε για οποιαδήποτε επιχείρηση, ξέρουμε ότι αν αυτό που θέλει κάποιος ε, είναι να χάσει ε, ουσιαστικά την επιρροή του ε, ή μερίδιο της αγοράς, τότε αλλάζει το όνομα. Ένα σοβαρός οργανισμός, καθώς ήδη λήφθη απόφαση να, να ονομαστεί έτσι ο οργανισμός, είναι σημαντικό να διατηρήσει το όνομά του. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή και μεγαλύτερες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια των δικτύων. Επίσης δεν συμφωνούμε με το να αλλάξει η έδρα του οργανισμού να φύγει από την Ελλάδα. Υποστηρίζουμε ότι όλα τα κρατημέλη πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά στο να έχουν στην επικρατεία του ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έτσι λοιπόν εγώ δεν ε, καταλαβαίνω γιατί η υπηρεσία αρμόδια για το περιβάλλον θα είναι στη Δανία και η ΕΝΙΣΑ δεν μπορεί να έχει έδρα στην Ελλάδα. Δεν συμφωνούμε λοιπόν να τροποποιηθεί η έδρα, να αλλάξει η έδρα. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να εισαγαγούμε μία σειρά κριτηρίων αποδοτικότητας, ίσως θα μπορούσαμε και να τα επιβάλλουμε μάλιστα, αλλά δεν υποστηρίζουμε να φύγει από την Ελλάδα. Κατόπιν, παρουσίασα μία τροπολογία έτσι ώστε τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να τα διορίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Κομισιόν. Και έχω και άλλη τροπολογία, η οποία λέει ότι τα καθήκοντα του οργανισμού θα πρέπει να συμπληρώνονται από ε, τη δράση των κρατών μελών ε, και η Κομισιόν φυσικά θα πρέπει να εκπονεί την κατάλληλη νομοθεσία για την ασφάλεια των δικτύων ε, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ικανότητας των κρατών μελών για να μπορούν να αποκριθούν σε ατυχήματα όταν έχουμε παραβίαση της ασφαλείας των δικτύων και επίσης να υπάρχουν και ομάδες προκειμένου να διευκολύνει το διάλογος, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αλλά και ακαδημαϊκών. Και κλείνω λέγοντας ότι η ασφάλεια των δικτύων ε, είναι κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο και πολύ σημαντικό εν ώψη του μέλλοντος. Και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα ισχυρό οργανισμό, μια ισχυρή ενίσα που να έχει και μια εντολή χωρίς χρονικό περιορισμό και επίσης υποστηρίζω να μείνει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο σκιώδεις ε, ζητούν το λόγο και μετά έχω έξι παρεμβάσεις. Παρακαλώ πολύ, ε, συντομεύετε, υπάρχουν και άλλα θέματα στην ημερήσια διαδέξη. Κυρία Βαλεάν. Um, Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον συγκητή για το έργο του, για την εκπόνηση της έκθεσης και επίσης ε, να τονίσω ότι η συνεδρίαση των σχεδόν ε, εισηγητών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για καρποφόρος. Όμως νομίζω ότι θα χρειαστούν ε, και άλλες συνεδρίσεις των σχεδόν ε, αφού είδα τις τροπολογίες, αν θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε συμβιβασμό γιατί στην έκθεση αυτή πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς βλέπουμε το μέλλον αυτού του οργανισμού. Καταρχήν, ε, να σας πω δύο λόγια για την έδρα. Δεν ε, είναι σημαντική η έδρα ή δεν είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, ε, όπως φαίνεται, αλλά υπάρχουν αρκετοί λόγοι να το λάβουμε αυτό υπόψη. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τοποθετηθεί για την έδρα, να θέλουμε να σεβόμαστε τις συνθήκες, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε μέσω αυτής της έκθεσης, να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο, προκειμένου να ξανασυζητήσει το θέμα της έδρας του οργανισμού. Δεύτερον, για τη διάρκεια της εντολής της ΕΝΗΣΑ. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των εισηγητών ε, επιθυμούν να υποστηρίξουν την ε, ιδέα να έχει μόνιμη εντολή ο οργανισμός. Και αυτό έχει φυσικά κάποια πλεονεκτήματα, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να έχουν καλή διαδρομία ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία σε αυτό το τομέα και θα συνεχιστεί προς το αξία των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Έτσι λοιπόν είμαι υπέρ της μόνιμης εντολής. Ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο. Νομίζω ότι το καθήκον αυτό θα πρέπει να το αναλάβει ο οργανισμός, να έχει νέα, νέους τομείς δραστηριοτήτων σε αυτή την εντολή για πολλούς λόγους ε, που ήδη αναφέρθηκαν από κάποιους συναδέλφους. Αλλά δεν νομίζω ότι ο οργανισμός θα πρέπει να γίνει ομάδα πληροφορικής άμεσης επέμβασης, ΣΕΡΤ, και ε, νομίζω ότι πρέπει να, να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα θα μπορούσε ο οργανισμός να έχει ένα χρήσιμο ρόλο ε, συνδεόμενη με τις διάφορες άλλες υπηρεσίες, με τους διάφορους άλλους οργανισμούς στον τομέα και εντοπίζοντας τα προβλήματα και τις τάσεις ε, και δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα και μόνο σημείο επαφής ε, για τις ε, τρίτες χώρες, ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, γιατί αυτό θα υποσκάψει την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών των διοκτικών αρχών. Σε ό,τι αφορά στην προστασία των δεδομένων, πιστεύω ότι η ΕΝΙΣΑ θα πρέπει να διαμετρήσει ένα ρόλο ε, στο να επικοινωνεί με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τις ε, εθνικές αρχές ε, πληροφοριών. Προτείνεται να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες ό,τι αφορά τις γνωμοδοτήσεις και τις αναλύσεις που θα εκπονεί αντί να βασίζεται μόνο στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν και να περιμένει να ζητήσουν αυτά τέτοιες αναλύσεις. Θα πρέπει η να έχει περισσότερη πρωτοβουλία δηλαδή. Και νομίζω λοιπόν ότι εδώ ένα σημείο καμπή για την Ενίσα και δεν θα ήθελα να διατηρήσω έναν οργανισμό που δεν θα έχει του κατάλληλου πόρου. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί λοιπόν για το θέμα αυτό, θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό αυτό με του απαιτούμενου πόρου. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Και να συγχαρώ τον Τζάιλς Τσίτσεστερ για την εξαιρετική δουλειά ε, και για την αφοσίωση που έχει δείξει σε αυτό το θέμα. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι έχω καλυφθεί αρκετά με αυτά τα οποία έχουν αλεχθεί και ιδιαίτερα από αυτά τα οποία είπε η κυρία Τικάου, που συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε. Επαναλαμβάνω ότι από πλευράς μας θα θέλαμε μία διεύρυνση και επέκταση του ρόλου της ΕΝΗΣΑ. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να αλλάξει το όνομα. Το branding υπάρχει, εκτός αν η αλλαγή του ονόματος υπενήσεται και κάτι άλλο, ε, το οποίο δεν μπορώ πράγματι να το καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να γίνει. Ε, την Ενίσα την βλέπουμε να έχει και επιχειρησιακό χαρακτήρα και επίσης να διευρύνει θα πρέπει να εκ των ε, ουκάνευ τη διεθνή τη συνεργασία ε, με άλλους οργανισμούς διεθνώς. Αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι θα θέλαμε η εντολή να έχει μόνιμο χαρακτήρα γιατί αν δεν έχει και δίνει μία διάρκεια 5 έως 7 ετών πάλι αυτό δίνει μία προσωρινότητα στο περιεχόμενο της εργασίας το οποίο θα γίνεται και οι εργαζόμενοι εκεί θα αισθάνονται ότι είναι προσωρινοί. Θα έλεγα λοιπόν ότι εισηγούμαστε να υπάρχει ένας μόνιμος χαρακτήρας ε, στην εντολή. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την αλλαγή της ε, ε, του Βένιου οπωσδήποτε δεν συμφωνώ. Αν ξεκινήσουμε από την Ελλάδα, μετά η μισή Ευρώπη ή τα δύο τρίτα της Ευρώπης θα πρέπει να μεταφέρουν όλους τους περιφερειακούς οργανισμούς. Αν υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα, θα πρέπει να τα δούμε και να δούμε τι λύση θα μπορούσαμε να δώσουμε, αλλά τα σοβαρά αυτά επιχειρήματα μέχρι τώρα δεν τα έχω ακούσει. Οπότε παραμένουμε και επιμένουμε στην παραμονή της έδρας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όλοι οι σκιώδεις της ομάδας μίλησαν, τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις. Έξι είναι. Προτείνω να περιορίσουμε το χρόνο ομιλία στα δύο λεπτά για να προλάβουμε. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά να προλάβουν όλοι. Η κυρία Αντεκαστήγια είναι η πρώτη. Eh, Μάλιστα, πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε λιγότερο από δύο λεπτά. Δεν θα επαναλάβω κανένα επιχείρημα, ούτε ε, θα συζητήσω επί των επιχειρημάτων που παρουσιάσαμε τροπολογίε, νομίζω ότι μπορούμε να τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε ως κύριο στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά την επιτέλεση των καθηκόντων και των στόχων ε, ενός τέτοιου οργανισμού. Οι τεχνολογίες ε, πληροφορικής έχουν ε, εξελιχθεί πάρα πολύ και επομένως η απάντηση που πρέπει να δοθεί τώρα δεν σχετίζεται μόνο με τις ελλείψεις και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, αλλά και με τις νέες αναγκαιότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή που δημιουργήθηκε ο οργανισμός. Λευθέντως αυτού δεν νομίζω ότι το θέμα της έδρας ε, ε, θα γίνει ένα θέμα που θα πολλώσει τη συζήτηση, γιατί διαφορετικά ε, δεν θα μπορούσαμε να βγούμε πολύ εύκολα από μια τέτοια κατάσταση, γιατί θα ήμασταν όλοι πολύ συναισθηματικοί απέναντι στο θέμα. Εγώ Νομίζω ότι αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειες στην αποτελεσματικότητα και να έχουμε κάποιες μόνιμες επαφές με ευρωπαϊκά όργανα, με άλλους φορείς, με τα κράτη-μέλη κτλ, ο οργανισμός και θα είναι μόνη περίπτωση, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γραφείο στις Βρυξέλλες ε, και μάλιστα ένα μεγάλο γραφείο. Εγώ νομίζω ότι έτσι μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα. Αυτά από μένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ υποχρεωτικά σύντομος. Άκουσα τους συναδέλφους, πολλοί από αυτούς με κάλυψαν. Θέλω μερικά σημεία να σημειώσω. Καταρχήν υποστηρίζω ότι ο ΕΝΙΖΑ είναι από τους μικρότερους οργανισμούς της Ευρώπης. Αποτελείται από 60 ανθρώπους και έχει προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν για cyber security η Βρετανία εξοδεύει 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει αυξημένο διεθνή ρόλο και αυξημένη ορατότητα, τόσο σε σχέση με διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται σε θέματα διαδικτύου, όσο και με τους διεθνείς μας εταίρους. Άκουσα με έκπληξη τις απόψεις του κυρίου Τσίτσεστερ σχετικά με το πώς γίνεται πώς λειτουργεί ένας οργανισμός που έχει καθήκον να εξασφαλίσει την cyber security. Τον άκουσα να μιλάει με υποτιμητικό τρόπο για την δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε με video conference ή με Skype. Υποθέτω ότι δεν έχει ακούσει και το Eurogroup και Summit γίνονται με αυτές τις μεθόδους και ίσως θα μπορούσε να έχει τη χρήσιμη πληροφορία ότι μόλις πρόσφατα το Αμερικανικό Κογκρέσο με Skype εργάζεται με σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας αλλά και των δαπανών. Ο κύριος Τσίζεστερ κατέθεσε μία έκθεση, το πρώτο μέρος της οποίας έχει να κάνει με την προτάσεις του για την ενίσχυση του ΕΝΙΖΑ, τη βελτίωση της διοικητικής του δομής και την αποτελεσματικότητά του, στον οποίο καταθέτει αρκετές θετικές προτάσεις πάνω στις οποίες εμείς έχουμε επίσης συμβάλει με δικές μας τροπολογίες. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την προσωπική του αντίληψη, την οποία είχε διαμορφώσει ήδη από την πρώτη επίσκεψη στον Ενίζα 18 μήνες από την ίδρυσή του και που έχει να κάνει με την απομάκρυνση του Ενίζα από το Ηράκλειο. Ένα λογικό τρίκ γίνεται εδώ. Αλλάζουμε τον στόχο, αλλάζουμε το όνομα και αλλάζουμε την έδρα. Όμως ε, κύριε Πρόεδρε, θα υποστηρίξω με τεχνοκρατικούς όρους και θα ενημερώσω τα μέλη της Ήτρας με, με εκτενέστερο κείμενο ότι η έδρα του Ηρακλείου δεν είναι απλώς επειδή το Ηράκλειο είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά διότι έχει όλες τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για να υποστηρίξει τον ενισχυμένο ρόλο του ΕΝΙΖΑ. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι αδιανόητο στην εποχή μας η κοζερή των υπαλλήλων μεταξύ των ομολόγων τους να χρειάζεται ε, μετακινήσεις τόσο συχνές όσο λέει. Οι εκθέσει του κυρίου ΟΣΥ δεν λένε τέτοιο πράγμα από το κόρτο και νομίζω ότι μια πιο εκτεταμένη συζήτηση που θα συμπεριλάμβανε και το satisfaction, το staff satisfaction report που βλέπω ότι δεν είναι ακόμα εις γνώση της Ήτρε θα ήταν μόνο ότι έχει κυκλοφορήσει από τον Ιούνιο θα βοηθούσε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανίστελ ε, Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να αντιδράσω και εγώ σύντομα. Νομίζω ότι ανέφερε κάποια ζητήματα ο κύριος Τσίτσεστερ, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή δυνατότητα του οργανισμού. Ο ΕΝΙΖΑ, υπό την παρούσα του δομή, ανταποκρίνεται σε, στις προσδοκίες και σε ό,τι αφορά την πολιτική συζήτηση και σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των κρατών μελών. Υπάρχουν αμφιβολίες. Εκπονείται μια έκθεση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το Critical Information Protection. Εγώ είμαι σκιώδης συζητητής για την έκθεση αυτή. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι σε τέτοιου είδους συζητήσεις ε, πάντοτε καταλήγουμε στην ευχή σύστασης νέων δομών και ενίσχυσης της συνεργασίας ε, σε κοινοτικό επίπεδο έχουμε λοιπόν ε, προτάσεις για μια σειρά πρωτοβουλίες για την διεθνή συνεργασία. Σε επαγρυπνήσουμε λοιπόν γιατί αν ο ΕΝΙΖΑ παραμείνει ε, με την ισχύουσα βάση, μήπως ε, τελικά και σε, άλλες, σε άλλους οργανισμούς ε, δημιουργηθεί πρόβλημα με τις δραστηριότητες που θα ροκανίσει σιγά σιγά ο ΕΝΙΖΑ. Όπως υπόθηκε υπάρχουν συζητήσεις και θα ακούσουμε επικρίσεις και κριτική και στο μέλλον. Δεν θέλω τώρα να αποφανθούμε ευθύ αμέσω για το θέμα της έδρας, αλλά σίγουρα πρέπει να το συζητήσουμε και σίγουρα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο ε, αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. You use it or you lose it. Αυτό είναι το δικό μου σλόγγαν και νομίζω ότι αυτό είναι και το αποφασιστική σημασία στοιχείο. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τα τοπικά συμφέροντα αλλά και τα ευρωπαϊκά. Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα δεν είναι τρομερή, άρα δεν θα έπρεπε να παραμείνει ως έχει οργανισμός. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τσίτσεστερ για την έκθεσή του. Θα ήθελα επίσης ε, να συγχαρώ και τους σκιώδεις εισηγητές ε, για τη δουλειά τους. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα έχουν ήδη υποθεί, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας όπως άλλωστε έκανε και ο προλαλής σας κύριος Νίστελ Ρόι, ε, στο, στις σοβαρές διαστάσεις που τίνει να προσλαμβάνει η κυβερνοασφάλεια ε, σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει ναι μεν να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται από αυτό φόρο, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιοι προληπτικοί μηχανισμοί για να μην υπάρχουν αυτού του είδους ε, οι δράσει και θα πρέπει να υπάρξει η διεθνή συνεργασία, η ευρωπαϊκή συνεργασία για να έχουμε πρόληψη, αποτελεσματική πρόληψη. Ξανασυζητούμε τώρα την εντολή του οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ο ρόλο του, δηλαδή να συντονίζει τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον ρόλο αυτό θα πρέπει να τον ενισχύσουμε και θα πρέπει να του δώσουμε και μία ε, εντολή ε, είναι ε, δυνατό να γίνει ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς αυτός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης της σημασίας που μπορεί να προσλάβουν οι επιθέσεις στον χώρο. Το θέμα της έδρας θα έλεγα να λυθεί ως εξής, να παραμείνει έδρα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος ε, έχει να κάνει ε, με τις τεχνολογίες, άρα μπορούσε να έχει την έδρα του οπουδήποτε στην Ευρώπη για να μην πω και στον κόσμο, ακριβώς αφού χρησιμοποιεί ως ε, βασικό το εργαλείο το διαδίκτυο οι ειδικοί του ΕΝΙΖΑ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίρνουν τις βάλτσες τους και τους χαρτοφυλακές τους στο χέρι και να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο αφού μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης δεν νομίζω ότι πρέπει να μετονομαστεί ο οργανισμός. Μόνο αν έχει αμαυρωθεί το όνομα κάποιου το αλλάζει κάποιο φορέα. Αλλιώς γιατί να αλλάξει. Κύριο Σοντή, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σε συνέχεια ε, της εξαιρετικής παρέμβασης του συναδέλφου Έλερ θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις καταρχάς ό,τι αφορά τη διάρκεια της εντολής ή μάλλον πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Όλοι οι συμπολίτε μας επιθυμούν την ασφάλεια, την οικονομική, τη λογιστική, τη σωματική ηλική ασφάλεια, την ε, άμυνα. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της έντολη, υπάρχει μια τροπολογία για ε, να περάσει από 5 σε 7 χρόνια η εντολή. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι θα πρέπει επαόριστο να ισχύει η εντολή του οργανισμού Αλλιώς ε, ίσως δεν έχει καν νόημα να υπάρχει αυτός ο οργανισμός αν δεν έχει αόριστη εντολή. Τώρα θα πρέπει να υπάγεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που δεν έχουν ενοποιηθεί στους ε, λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο συγκεκριμένος οργανισμός υπάγεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον από αυτήν ορίζονται οι εργαζόμενοι σε αυτόν και θα πρέπει να υπάρχει ίσως ε, μια ποσόστοση διοικητικών υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς πτυχές, η τροπολογία 117 για το άρθρο 28 προβλέπει ότι ο οργανισμός ε, θα μπορούσε να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αυτό θα ήταν σοβαρό σφάλμα. Ο οργανισμός πρέπει να υπόκειται και στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν θα πρέπει να συναλλάσσεται με χώρες στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών χωρίς αυτό να πλαισιώνεται από την Ένωση. Και μία τελευταία λέξη για την έδρα. Ο ε, κύριος ε, Τσίτσεστερ μας έχει συνηθίσει σε επίδειξη ανοιχτού πνεύματος. Είπε ότι δεν θα είναι δημοφιλή στην Ελλάδα με κάθε ειλικρίνεια, ε, νομίζω το μόνο που τον ενδιαφέρει να είναι δημοφιλή στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι η επίθεση αυτή κατά τη έδρα δεν είναι στο ύψο ε, όσων διακυβεύονται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχουμε κατανείμει τι έδρε ουσιαστικά, γιατί θέλαμε να υπάρχει ε, συγχρονισμό ενό επιμηξία, θα έλεγα, των διαφόρων υπαλλήλων. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Παραδείγματο χάρη με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράγκμπι στη Νέα Ζηλανδία, κύριε Τσίστερ, είστε και μέλο ε, της ε, αντιπροσωπείας με την Νότια Αφρική και την ε, Νέα Ζηλανδία. Τι πρέπει να κάνουμε, τα σταματήσουμε όλα στον κόσμο. Λοιπόν, εγώ στηρίζω τον κανόνα της κατανομής των εδρών. Θα δούμε αν σε 10-20 χρόνια αν θα πρέπει να έχουμε μια ομόσπονδη πρωτεύουσα. Είναι πολύ εύθραυστη όμως σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη για να σταματήσουμε αυτήν την επιμειξία, αν θέλετε, αυτό το συγχρονισμό των υπαλλήλων των διαφορετικών χωρών της Ένωσης. Κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω το σημείο της ε, σύνδεσης της αποδοτικότητας με την έδρα του οργανισμού. Φυσικά θέλουμε αποδοτικότητα, αλλά θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τα δύο αυτά ζητήματα. Και όπως είπε και ο κύριος Σοντή, Υπάρχει μια ολοκλήρη φιλοσοφία ε, που διέπει την κατανομή των ε, εδρών των ευρωπαϊκών οργάνων ε, και θέλω να αναφερθώ στον ε, πρόεδρο Σαρκοζή όταν ε, ε ξεκινάει η συζήτηση ε, για τους, ε, τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, ε, αν αρχίσουμε να συζητάμε εδώ το θέμα των εδρών, θα πρέπει να συζητήσουμε τα πάντα και για τις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΕΚΤ και τα λοιπά, γιατί υπάρχει τώρα μια φιλοσοφία ισορροπία στη γεωγραφική κατανομή και δεν θα πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αποδοτικότητα αυτού του οργανισμού, χωρίς το στάδιο αυτό να αμφισβητούμε το θέμα της έδρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και η συνάδελφος κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ λεπτό. Διαδικαστική παρατήρηση από τον κύριο Οντί. Συγγνώμη, κατόπιν την παρέμβαση στις συναδέλφους, ίσως να υπήρχε ένα πρόβλημα στη μετάφραση. Να πω ότι δεν υπάρχουν δύο έδρες. Ε, η έδρα είναι στο Στρασβούργο, απλώς έχουμε τρεις τόπους εργασίας. Κύριε Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη γιατί έχω καλυφθεί από αρκετούς συναδέλφους που μίλησαν νωρίτερα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτά στα οποία συμφωνούμε σε ό,τι αφορά στον ΕΝΙΖΑ. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τον οργανισμό αυτό Συμφωνούμε ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τη διοικητική του δομή και την αποτελεσματικότητά του. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να παραμείνει ο οργανισμός ως έχει. Θέλουμε όλοι αλλαγές. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να τον αναβαθμίσουμε αυτόν τον οργανισμό, να βελτιώσουμε τη λειτουργία του, να αξιολογήσουμε την εντολή του και ως, προς το περιεχόμενο και ως προς τη διάρκεια, να δούμε δηλαδή αν αυτή η περιορισμένης διάρκειας εντολή που έχει ο οργανισμός αυτό σήμερα είναι συμβατή, συνάδει με το περιεχόμενο της εργασίας αυτού του οργανισμού, με τους στόχους του και αν δίνει επαρκές κίνητρο στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στο επιστημονικό προσωπικό, για το οποίο τόσα λέγονται και τόσο πολύ ενδιαφερόμαστε και πολύ σωστά, για να κάνει καριέρα σε έναν τέτοιον οργανισμό. Να κάνει καριέρα σε έναν τέτοιο οργανισμό εφόσον έχει προοπτική. Η αλλαγή ονόματος όμως, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η συνεπακόλουθη, διότι συνδέονται αυτά τα δύο κατά τη γνώμη μου αλλαγή έδρας, δεν μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν τα προαναφερόμενα, η αναβάθμιση του οργανισμού, η αξιολόγηση της εντολής του, του περιεχομένου της εργασίας του. Πρώτα απ' όλα διότι σήμερα, όπως πολύ σωστά είπε η ε, συνάδελφος πριν, οι ανάγκε σήμερα έχουν αλλάξει και οι τεχνολογίε εξελίσσονται και το υπενθύμησε και ο κύριο Τσουκαλά στην παρέμβασή του, η εξέλιξη των τεχνολογιών ακριβώς αποδυναμώνει το επιχείρημα τη ισχύω τη έδρα σε ό,τι αφορά τι λειτουργίε αυτού του οργανισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνολογικά μέσα σήμερα στη διάθεσή μα, ε, που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε εξαιρετική δουλειά εξ αποστάσεως και αυτό το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν λέω ότι είναι σωστό ότι δεν πρέπει ε, να επικεντρωνόμαστε, κάποιος συνάδελφος το είπε, στα τοπικά συμφέροντα. Υπάρχει το ευρωπαϊκό συμφέρον. Από την άλλη, ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε ως άλοθη επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με την ουσιαστική λειτουργία του οργανισμού για να ανοίξουμε θέματα, να ανοίξουμε το μοναδικό θέμα στην πραγματικότητα, που μεθοδεύεται εδώ και αρκετό καιρό και που αφορά στην αλλαγή της έδρας του οργανισμού. Όταν αποφασίσαμε, όχι μόνο για τον Εμίζα, η λογική που διέπει τα κριτήρια στα, με βάση τα οποία έχουμε συμφωνήσει ότι επιλέγουμε τις έδρες των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών, που είναι μια λογική αποκέντρωσης απαντούσε και απαντά σε ορισμένα επιχειρήματα. Κυρίως το γεγονός ότι δεν θέλουμε να περάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι μόνο οι Βρυξέλλες και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ παλιότερα, είναι μόνο οι κεντροευρωπαϊκές χώρες. Θέλαμε ακριβώς να περάσουμε το μήνυμα και θέλουμε πιστεύω να περάσουμε το μήνυμα παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα ότι η Ευρώπη είναι και αποκέντρωση και ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα περισσότερο όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ασφαλώς, αλλά και τα ίδια δικαιώματα. Δεν είναι οι περιοχές αυτές, ούτε οι πολίτες των χωρών αυτών, περιοχές και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για να κλείσω λοιπόν, είναι σαφές ότι θα πρέπει και συμφωνώ απολύτως να προτάσουμε το ευρωπαϊκό συμφέρον στην αξιολόγησή μας. Δεν πρέπει να επικρατούν τοπικά κριτήρια, κριτήρια τοπικού συμφέροντος. Ταυτοχρόνως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει αντιστοίχως σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που περνάμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να χρησιμοποιούμε κατά κάποιο τρόπο τις δυσκολίες αυτής της κρίσης για να μεθοδεύσουμε ε, από το παράθυρο ε, αιτήματα τέτοιου τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Προεδρίας, ο κύριος Ματσίνσκι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, Είναι τιμή μου που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση και η Πολωνική Προεδρία αλλά και άλλα κράτη-μέλη. Περιμένουν με ανυπομονησία την έκθεση αυτή και φυσικά αναμένουμε με ανυπομονησία και την έγκρισή τη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συντάκτη τη έκθεση, τον κύριο Τσίτσεστερ και του συνεργάτε του. Πιστεύουμε ότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας ε, των δικτύων μας ICT. Η Πολωνική Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει ένα πολιτικό συμβιβασμό και θα προσπαθήσει να υιοθετήσει τον κανονισμό εμείς ε, συμφωνούμε ότι η εντολή του οργανισμού θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη. Θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ασφάλεια των τεχνολογιών ε, πληροφοριών και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς που καλύπτουν την ασφάλεια στο διαδίκτυο και θα πρέπει να έχει και τους καταλληλούς δημοσιονομικούς πόρους. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές προκλήσεις ε, στην εργασία μας και θέλουμε μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και με το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Είδαμε πολύ καλή θέληση και είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Επίσης, ευχαριστούμε και τον κύριο Τσίτσεστερ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές στις ε, εργασίες μας και ελπίζουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Η υιοθέτηση αυτού του κανονισμού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πρόκειται για μια απόφαση που ε, την περιμένουν εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου. Η κυρία Αντζελόβα από την Κομισιόν, ελπίζω να το λέω σωστά, η κυρία Αντζελόβα ή ποιος άλλαξε. Ε, ευχαριστώ. Η ποιος αλλαξε πρότεινε νέα εντολή για τον ΕΝΙΖΑ θεωρώντας ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός και ενίσχυση της εντολής του ΕΝΙΖΑ. Μια σημαντική πτυχή ήταν η πενταετής διάρκεια της θητείας. Γιατί η Κομισιόν θεωρεί ότι οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα είναι τόσο ραγδαίες, ώστε χρειάζεται σε τακτά διαστήματα μια αξιολόγηση σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η πρόταση είναι καλή βάση για τις ε, συζητήσεις για τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση του ΕΝΙΖΑ όπως λέει το Κοινοβούλιο, όπως θέλει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την έκθεση και παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την σχετική συζήτηση στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Τέλος, ο κύριος Τσίτσεστερ για να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα πολύ επικοδομητικά και χρήσιμα σχόλια και τη συζήτηση. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία του Συμβουλίου σήμερα εδώ και ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις ευγενικές παρατηρήσεις αναφέρω το Συμβούλιο γιατί δείχνει ότι αναγνωρίζουν τη σημασία του θέματος και της συζήτησης. Ευχαριστώ. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα μετά τα σχόλια των συναδέλφων. Καταρχήν, το ζήτημα της αλλαγής ονόματος και έδρας αλλαγής. Ως συντηρητικός θεωρώ ότι είναι μια ηρωνία το γεγονός ότι οι συνάδελφοι εξ αριστερών παρουσιάζονται συντηρητικοί, μη αποδεχόμενοι την αλλαγή, ενώ εγώ συντηρητικός θέλω την αλλαγή. Υπάρχει εδώ μια πολύ ευχάριστη ηρωνία. Πέραν τούτου, σε εύθετο χρόνο θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση ε, στην ευρωπαϊκή αυτή προσέγγιση. Έγινε μια παρατήρηση σχετικά με το ζήτημα της έδρας ότι δηλαδή ο οργανισμός περιβάλλοντος μπορεί να είναι στη Δανία. Γιατί ο ΕΝΙΣΑ λοιπόν να μην είναι στην Ελλάδα. Αυτές και οι δύο είναι πολιτικές αποφάσεις. Όμως ε, η γεωγραφική κατάσταση διαφέρει γιατί η Δανία είναι λίγο πιο κοντά στην καρδιά της Ευρώπης. Δεύτερον, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ότι ο οργανισμός θα έπρεπε να πάει στην Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν για την Κρήτη. Και εδώ έχουμε γεωγραφική διαφορά, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Είναι αντικειμενικό αυτό. Τώρα, η διάρκεια της θητείας. Η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να είναι πενταετής η θητεία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσω με την σύσταση της μελέτης και της έκθεσης που κατατέθηκε και είναι καλά τεκμηριωμένη και καλογραμμένη η μελέτη αυτή και λέει ότι υπάρχει μια λογική στο να συμπίπτει με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές η θητεία. Οπότε πρέπει να είναι επταετής η θητεία. Μπορούμε να πούμε και για όριστη ε, σε χρόνο, σε διάρκεια ε, εντολή, αλλά πώς ξέρουμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 100 χρόνια, το ξέρουμε. Όχι, θα έλεγα εγώ. Αν είναι επαόριστον η θητεία θα πρέπει να προβλέψουμε τακτές αξιολογήσεις ανά πέντε χρόνια για να κρίνεται η αποτελεσματικότητα και η αξία του οργανισμού. Είναι τρίτη φορά από ό,τι γνωρίζω που το κάνουμε αυτό στην ε, σύντομη ζωή αυτού του οργανισμού. Γιατί, Γιατί είμαστε σε ένα τομέα τεχνολογίας και πραγματογνωμοσύνης που αλλάζει ταχύτατα και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το λάβουμε υπόψη και να συμμορφωθούμε προς αυτό το δεδομένο. Η επταετής θητεία δεν σημαίνει ότι περιορίζεται εκεί. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 7 χρόνια θα χρειαστεί να ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση ή μη όχι. Και για ποιο λόγο. Και αυτό κάνουμε μετά από 7 ή 8 χρόνια. Αυτό κάνουμε τώρα, 7-8 χρόνια μετά τη σύσταση του οργανισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι λογικό και δεν πιστεύω ότι ε, αν πούμε ότι ε, θα είναι επταετής. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια στους απασχολουμένους στον οργανισμό. Απογοητεύτηκα λίγο που η συνάδελφος κυρία Τζαβέλα, που τη σέβομαι ιδιαίτερα για τις διανοητικές της ικανότητες, είπε ότι δεν άκουσε σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής της έδρας. Εγώ νόμιζα ότι είχα δώσει πολύ σοβαρά επιχειρήματα για την αλλαγή. Αλλά θα έπρεπε να πω, για να αντικρούσω, ότι δεν άκουσα σοβαρά επιχειρήματα υπέρ του Ηρακλείου καταρχήν. Εκτός από το ότι θα έπρεπε πούμε, η τοπική οικονομία μιας περιφέρειας να υποστηριχθεί. Για να το δούμε λίγο. Φαντάζομαι ότι κάποια λύση υπάρχει, πάλι ε, πάνω στη βάση του συμβιβασμού. Μπορεί να μην συμφωνήσετε μαζί μου σχετικά με την έδρα και εγώ μπορεί να μην συμφωνήσω μαζί σας. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα βρούμε μια λύση ενδιάμεση. Επίσης, για να αναφερθώ στα όσα είπε ο κ. Τσουκαλάς. Και χαίρομαι που είχαμε τόσες ελληνικές παρεμβάσεις, ε, γιατί εγώ τώρα είμαι λίγο σαν outsider σε αυτή τη μικρή λέσχη την ελληνική. Είπε ότι είναι αδιανόητο ε, να χρειάζεται να πηγαίνουν έρχονται οι συνεργάτες. Μα πρέπει όμως, γιατί πρέπει να συναντούν ο ένας τον άλλον. Εσείς ε, μπορεί να λέτε ότι δεν είναι σωστή η προσέγγιση μου υπέρ των τηλεδιασκέψεων. Είναι άδικο όμως αυτό. Νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η προσωπική επαφή. Και είναι σαφές από αυτά που κάνουν τώρα και σας παραπέμπω στη μελέτη και πάλι ότι πραγματικά γίνονται πάρα πολλά ταξίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του οργανισμού. Χαίρομαι διότι τα επιχειρήματα όλα τάσσονται υπέρ της μεγαλύτερης ε, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας του οργανισμού. Νομίζω ότι όλοι δέχονται ότι θα πρέπει ο οργανισμός να ασχολείται περισσότερο με την ασφάλεια του διαδικτύου και την ασφάλεια των δικτύων, πολύ περισσότερο από ότι ε, τα διοικητικά, γιατί το διοικητικό κομμάτι δεν είναι μόνο η ουρά του οργανισμού, αλλά έχει φτάσει να είναι και το κεφάλι. Πρέπει να αντιστραφεί η σχέση δεν, ε, η κυρία Τίκαου μίλησε για κάποιες αναλογίες. Δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ απόλυτα, αλλά κάτι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ όλους για τις επικοδομητικές παρατηρήσεις και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις, όποτε θα έχουμε την ευκαιρία να ε, επεξεργαστούμε και να μελετήσουμε τις τροπολογίες και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε διαδικαστική παρέμβαση του κυρίου Τσουκαλά. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι η κατανομή του χρόνου ομιλίας είναι άνηση. Αν το διαφέρομενο μέρος ε, από τη μία πλευρά έχει πολύ χρόνο να μιλήσει και στη συνέχεια εμείς περιοριζόμαστε στα δύο λεπτά. Εγώ το σεβάστηκα απόλυτα αυτό το χρονικό όριο. Δεν, τότε στη συνέχεια δεν μπορώ να πω ότι για τεχνικούς ε, λόγους, για ποιους τεχνικούς λόγους η έδρα πρέπει να είναι στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν ε, θα στείλω ένα αναλυτικό κείμενο στα μέλη της Επιτροπής Ήτρε και θα συμπεριλάβω τα όσα ήθελα να πω και δεν είχα χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση αυτή και την προσφορά. Πάντα έχουμε πρόβλημα χρόνου ε, και βέβαια δεν μπορεί κανείς να είναι πάντα δίκαιος στην κατανομή, αλλά μιλήσαμε ε, κατά μισή ώρα περισσότερο για αυτό το θέμα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Θέλαμε να ε, νοικοκυρέψουμε το χρόνο, να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στους σκιώδεις, νομίζω θα συμφωνήσετε με αυτό. Και μετά έδωσα σε όλους δύο λεπτά. Και κάποιοι συνάδελφοι τήρησαν το χρόνο, κάποιοι υπερέβησαν τα όρια, τα χρονικά που τους είχα δώσει. Παρακαλώ πολύ να ε, το λαμβάνουμε αυτό υπόψη ε, για να ε, μην χρειάζεται να διακόπτουμε. Παρακαλώ τώρα μην συνεχίσουμε με τα διαδικαστικά, γιατί δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε τα άλλα. Η κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Για να ενημερώσω εδώ τους συναδελφούς, το Ηράκλειο είναι ένας από τους ε, μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Danke für diesen Ευχαριστώ πολύ για αυτή την προσθήκη, σημαντική. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο σημείο ε, και θα ε, αναφερθούμε σε αυτό όπως είπε και ο κύριος Τσουκαλάστος στο προηγούμενο. Λοιπόν, αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κυρία Σαρτόριος, η συγγήτρια έχει το λόγο. Τώρα θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο ε, σε όλα τα σημεία μας. Κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Της 15 ε, Σεπτεμβρίου έστειλα την ομοδότηση στις μεταφραστικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, ε, είμαι στη διάθεση των συναδέλφων και επίσης ε, την ίδια ημέρα ε, κοινοποίησα στους σκιώδεις συζητητές, Ράμε Κορέντα και τα λοιπά, την πρόθεσή μου να έχω μια συνάντηση μαζί τους ε, την εβδομάδα της ενομέλίας Έτσι λοιπόν, ελπίζω ότι θα έχουμε την ε, δυνατότητα να έχουμε μια μεγαλύτερη ανταλλαγή απόψεων τότε. Γνωρίζουμε όλοι πόσο πολύ έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο το σχέδιο από την στιγμή της σύλληψής του και μένουμε για, έτσι ώστε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να έχει δική του γραμμή προπολογισμού. Το ΙΤΕΡ, όπως ξέρετε, μεταξύ του 2008 και του 2010 η οργάνωση ΙΤΕΡ έκανε μία ανάλυση του κόστους. Θα ήθελα να παρακαλέσω να σταματήσετε το χρόνο που τρέχει, γιατί υπάρχει φασαρία. Κοιτάξτε, μπορώ να μιλάω σε μια άδεια αίθουσα, αλλά όταν υπάρχει τόσο θόρυβος δεν μπορώ να μιλάω. Λοιπόν, όπως ε, γνωρίζετε, μεταξύ 2008 και 2010 ο οργανισμός Ήτερα έκανε μια ανάλυση του κόστους ε, προσπαθώντας να επικαιροποιήσει τις ε, χρηματοοικονομικές ανάγκες ε, του σχεδίου και ε, για διάφορους λόγους ε, προκαλύφθηκε ότι για να καλυφθούν διάφορες τεχνικές επιστημονικές και δικαιό... αναγκαιότητες και διαχείρισης του ΙΤΕΡ θα χρειαστεί επιπλέον προπολογισμό και στη συνέχεια πέρασε στο 1.300.000.000 εκατομμύρια και κατόπιν της εφαρμογής μία εσωτερικής πολιτικής συγκράτησης του κόστους σε σχέση με το αρχικό ποσό που είχε προβλεφθεί που ήταν 6,6 δισεκατομμύρια. Το Κοινοβούλιο ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει σε σχέση με τον τρόπο χορήγησης των πρόσθετων πόρων. Επανειλημμένα έχει εκφράσει την υποστήριξή του στο σχέδιο Ίντερ στο σύνολό του, στο έργο Ίντερ. Επίσης ε, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες όμως σε σχέση με τους τρόπους χρηματοδότησης πέρσι. Εκφράστηκαν ε, οι για την πρόσθετη χρηματοδότηση για το 2010 και εμείς σταθήκαμε υπέρ και υποστηρίξαμε ένα τμήμα των πόρων που βρίσκονται στο τομέα 1α, ανταγωνιστικότητα για την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη να δοθούν εκεί φέτος. Καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο για τα έτη 2012 και 2013. Η πρόταση της Επιτροπής σε με ανακοινώθηκαν σε άλλες περιπτώσεις και σε μεγάλο βαθμό τι συμμεριζόμαστε ε, πρόκειται για μια πρόταση που κινούταν σε δύο οδούς και η, ε, Κομισιόν διατήρησε τις υποχρεώσεις του Προτείνει αφενός ε, να ε, προσαρμόσει τον τομέα 2 ε, και τον τομέα 5 διοίκηση με για τον προπολογισμό του 2012 και 2013 φτάνοντας περίπου στα 840 εκατομμύρια ευρώ που θα ανακτηθούν. Από την άλλη προτείνει να δοθούει ένα τμήμα του υπολογισμού του 7ου προγράμματος, προγράμματος πλαισίου των ετών 2012-2013. Ως ε, εισηγήτρια για την Επιτροπή ε, δεν ήθελα εγώ να μπω στα ε, νούμερα. Εμείς... Ε, ε, δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουμε στις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις χρηματοδότησης ούτε την αρμοδιότητα. Εγώ αποφάσισα απλώ να κάνω το εξή να υπογραμμίσω αυτό ε, για το οποίο θεωρώ ότι είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν θα αποφασίσουμε επί της ουσίας και είμαι πεπισμένη ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα λάβει δεόντως υπόψη τις προτάσεις μας αφού έχουμε επαναλάβει την υποστήριξή μας ε, στο έργο ΙΤΕΡ και αφού ε, μελετήσαμε την ε, πρόταση της Κομισιόν, στη δεύτερη παραγράφο ήθελα να υπενθυμίσω ότι η χρήση του τομέα 1α δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλος γιατί Εκεί αυτός ο τομέας συμβάλλει σε μείζωνα βαθμό στους στόχους που θέτει η Ευρώπη 2020. Στην τρίτη παράγραφο απλώς ε, περιορίστηκα στο να εκφράσω την υποστήριξή μας ε, στη χρήση ενός μείγματος ε, χρηματοδοτικών πόρων περιλαμβανομένων και των διαθέσιμων περιθωρίων από τους διάφορους τομείς του σημερινού δημοσιονομικού πλαισίου. Στην τέταρτη παράγραφο αναφέρομαι στο ότι είμαστε αντίθετοι στην ε, χρήση των πιστώσεων του προπολογισμού από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για τα έτη 2012 και 2013. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο συμβάσει που έχουν ήδη συναντήσει και διαγωνισμούς που έχουν ήδη προβλεφθεί γιατί εδώ μιλάμε για τις δραστηριότητες του 7ου, του 7 προγράμματος πλαισίου μέχρι το 2013. Το Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει το θέμα αυτό και η ε, γνωμοδότηση που υθέτησε η δική μας Επιτροπή για τον προγραμματισμό του 2012 αναφέρει αυτή τη θέση. Στην παράγραφο 5 τονίζουμε την ε, ανάγκη να υπάρχει συγκράτηση του κόστους, να οργανωθεί ε, μια ε, διαχείριση ορθή και επακριβής χρηματοδοτικός σχεδιασμός και να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που γίνεται. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει πάντοτε να αξιολογούμε την πραγματική αναγκαιότητα της πρόσθετης χρηματοδότησης που ζητείτε και ε, κατόπιν ε, διάφορων πληροφοριών που μπορεί να επισέρχονται. Η τελευταία παράγραφος κατά την άποψή μου είναι σημαντική γιατί θα μας έδινε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στη διαδικασία και γραπτός στην περίπτωση που έχουμε σημαντικά νέα στοιχεία ε, και ε, ε, συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη του έργου ΙΤΕΡ. Αναφέρομαι στο σχέδιο προπολογισμού για το 2012 στο πρόγραμμα πλαίσιο σχετικό με την Ευρατομ ε, πριν πέθυνε για το 80% της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης και τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να υπάρχει μια γραμμή προπολογισμού που να αφιερώνεται στο έργο Ίτερ. ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, 18 Οκτωβρίου κατάθεση τροπολογιών ψηφοφορία στην Ήτρε 10 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Υπολογισμού το Νοέμβριο και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο του 2011. Ευχαριστώ. Ο Κορέρο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτόρη για αυτή την εξαιρετική έκθεση με την οποία συμφωνώ. γνωρίζουμε εδώ και καιρό το ύπαρξη του έργου Ίντερ και θεωρούμε ότι αποτελεί μια μελλοντική λύση για μελλοντικές ενεργειακές πηγές για την Ευρώπη. Έχει πολύ σημαντική προσθεμένη αξία, έχει εμβληματική σημασία και φέρει περιβαλλοντική αηφορία και επίσης έχει πάρα ε, πολλές σημαντικές συνέπειες σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη και αναφέρομαι ε, στην ενίσχυση των ικανοτήτων στη μηχανική των χωρών που συμμετέχουν ε, και πάντοτε πρέπει να έχουμε ε, κατά νου το πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτό. Είναι αλήθεια ότι τίθεται το θέμα του κόστους ε, και εμείς ε, πρέπει να κάνουμε εδώ κάποια χρηματοδοτική μηχανική για να καλύψουμε το κόστος αυτό. Συμφωνούμε με τις προτάσεις της ηγήτριας να αναζητήσουμε κάποιους πόρους από τους ίδιους πόρους και... Ε, να σας πω ότι δεν συμφωνούμε στο να αναζητήσουμε τους πόρους από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και συμφωνούμε εδώ με την εισηγήτρια δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συστάσεις της ηγήτριας θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον. Καταρχήν ε, πρέπει να αποφύγουμε αποκλήσεις ε, με μια καλύτερη διαχείριση και Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ίδιος προϋπολογισμός. Είναι πολύ θετικό η πρώτη πρόταση προϋπολογισμού της Κομισιόν να συμπεριλαμβάνει ξεχωριστά το ΙΤΕΡ από την χρηματοδότηση του 8ου προγράμματος πλαισίου και πρέπει να ασκήσουμε κάθε πίεση για να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στο Κανταράς με αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες για το ίτερ και σε ό,τι αφορά την κατασκευή πριν από κάποιες ημέρες, αν θυμάστε, είπε, η Ιαπωνία ότι θέλουμε δύο χρόνια για να τα ανταποκριθούμε στους στόχους. Άρα αβεβαιότητα. Άλλη αβεβαιότητα. Επιστημονικά προβλήματα που δεν έχουν επιληφθεί ακόμη και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή του ίτερ και ε, με ορίζοντα το 2100 ξέρετε ότι για τις προτεραιότητες έχουμε κάποια ζητήματα. Τα 1,3 δις πώς θα τα βρούμε από την έρευνα. Κοιτάξτε, η έρευνα έχει τις προτεραιότητές της, είναι ένας τομέας ε, αφεαυτού και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν από εκεί να προέλθουν οι πόροι. Επίσης, ό,τι αφορά ε, το έκτακτο κόστος, δεσμεύεστε ως Κομισιόν για τα επόμενα δύο χρόνια, ρωτώ, μιλάμε για το 2012-2013, δεσμεύεστε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος και αν υπάρξει ποιος θα το πληρώσει. Γιατί είμαστε τώρα σε μια κατάσταση, δεν ξέρω αν θυμάστε στην αρχή ήταν 4,7 δις, πέρασαμε στα 15 δις, εγώ θα ήθελα πραγματικά να γίνει μια πραγματική μελέτη επιπτώσεων. Δεν υπάρχει όμως μελέτη επιπτώσεων για το ζητούμενο ποσό και όλα αυτά βέβαια μαζί με τις αβεβαιότητες που υπάρχουν. Θα ήθελα λοιπόν να αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Μέζαρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτόρη για την έκθεσή της έκθεση στην οποία θέτει ζητήματα τα οποία αμφισβητούν ε, ή μάλλον θέτουν το πώς θα προχωρήσουμε με το ίτερ. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Θα ήθελα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πω ότι πολλοί θα ήθελαν ε, να θάψουν κάποια στιγμή το ίτερ. Εγώ σας λέω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Υπάρχουν ε, τα οικονομικά συμφέροντα αφενός, Έχουμε και την ενεργειακή ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια καθώς επίσης και για την εξασφάλιση ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητα, απαραίτητα μέσα και εργαλεία για αυτή την ενεργειακή ασφάλεια. Το ίτερ είναι μια δυνατότητα. Φυσικά και είναι ένα μακρόπνο έργο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ως πολιτικοί όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά και τα εγγόνια μας. σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ, τη μεγαλύτερη χρήση του, δεν νομίζω ότι αρκούν για να μα καλύψουν τι ενεργειακέ ανάγκε. Είμαστε σε μια εκθετική καμπύλη. Ε, Επομένω, ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε και τεχνικέ προκλήσει τεράστιε, όχι μόνο οικονομικέ. Αλλά αν υπερπηδήσουμε όλε αυτέ τι δυσκολίε, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη τεχνική επιτυχία. Στο Κανταράς έχω πάει και εγώ, θεωρώ ότι είναι βιώσιμο και νομίζω ότι καλό είναι να μην ε, κάνουμε βήματα προς τα πίσω και να μην ε, ε, φύγουμε από την θέση που έχουμε ως σκαπανή στον τομέα αυτό πρέπει να παροτρύνουμε να υπάρξει έρευνα και σε άλλα θέματα ε, που σχετίζονται με την ε, πυρηνική σύνδεξη. Έχουμε και τη σχάση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι ότι Πρόκειται και για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το πολιτικό κύρος και το πολιτικό γόητρο. Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με αυτό το έργο. Θα έπρεπε και η Ευρώπη να είναι αποφασισμένη να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση. Γιατί αλλιώς χώρες όπως είναι η Κίνα ή η Ρωσία ε, θα μας ε, προσπεράσουν ε, με γοργό βήμα. Αν δεν λάβουμε τις σωστές μας αποφάσεις το 2011, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και το 2012 και το 2013 δεν προβλέπονται επαρκή κονδύλια για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΙΤΕΡ. Είμαι κατά λοιπόν των προτάσεων της Κομισιόν. Νομίζω ότι πρέπει να ε, καλυφθούν ε, τα κονδύλια από το απόθεμα του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία του Air Καταρχήν, ε, δεύτερον, πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις ε, λόγω της επόμενης ε, συνάντησης ε, του Συμβουλίου και να σας πω ότι το σχέδιο JET είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σχέδιο σύντηξης. Ε, θέλω να υποστηρίξω την εισηγήτρια, τη χρήση των περιθωρίων και να μην χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, αυτό σημαίνει τα 460 εκατομμύρια λιγότερα για το 2012-2013, όμως ε, βλέπουμε ότι λόγω των προβλημάτων στην Ιαπωνία θα μπορούσε να αναβληθούν κάποια καθήκοντα. Έτσι λοιπόν δεν θα τίθεται σε κίνδυνο το έργο και θα έχουμε μια ισορροπημένη λύση. Υποστηρίζω λοιπόν τη λύση που προτείνει η συγγήτρια. Κύριε Σοντή, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγητριά μας ε, για το ισορροπημένο κείμενο. Και πάλι σημείωσα τις παρατηρήσεις σε σχέση με τους ε, κινδύνους ε, που αναφέρονται. Να πούμε ότι σήμερα σε μια κοινωνία χωρίς κινδύνους είναι αδύνατο, χωρίς ε, την ενέργεια της σύνδεξης. Να σας πω ότι Ξέρουμε καταρχήν ότι λειτουργεί, πρόκειται για ε, κάποιες εμπειρίες και κάποια πειράματα που ξεκίνησαν οι Ρώσοι. Έχουμε τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα, αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της ε, ε, και ταυτόχρονα είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να αποφύγουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά δύο βαθμούς. Τώρα, για τους τρόπους ε, χρηματοδότησης, απλώς να πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στις ε, δυσκολίες που έχουμε για τη χρηματοδότηση αυτού των μεγάλων έργων ε, που, χρήζουν, που χρειάζονται μεγάλα ποσά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το ίτερ χαίρομαι που η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ψήφισαν μια πρόταση για να δημιουργηθεί ένα τμήμα επενδύσεων, χρειάζεται ένα τέτοιο τμήμα επενδύσεων, ε, για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ευελιξία που μας προτείνεται εδώ, δηλαδή αν έχουμε πλεονάσματα ε, να μην τα δίνουμε στα κράτη-μέλη και να τα διατηρούμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να χρηματοδοτούμε τέτοια έργα μεγάλα κατά τα λοιπά. Υποστηρίζω την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη και νομίζω ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Και κάτι ακόμα πριν να μου αφαιρέσετε το λόγο, Πρόεδρε. Ε, να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν ε, έπλεξα παρκώς το κοινοβούλιο στις δυσκολίες Twitter. Ε, Τώρα αυτό έχει γίνει, αλλά δεν κατανοούμε πώς θα έχουμε μία πλήρη εικόνα για τη συνολική χρηματοδότηση του έργου. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστέρηση μισής ώρας και πρέπει να καλύψουμε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης που είχαμε και από την προηγούμενη φορά. Παρακαλώ λοιπόν σύντομα στις παρεμβάσεις, ίσως ενός λεπτού, ε, κυρία Χάρτσου, ε, η πρώτη από τους εννέα ομιλητές που έχουμε ακόμα. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύπτει ε, τα μεγάλα έργα και μεγάλες υποδομές. Πρέπει να ε, ορίσουμε τα μεγάλα έργα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για το ίτερ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια ως κοινοβούλιο δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο ελιγμών, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για το ίτερ, όπως είπε ο κύριος Όντι άλλωστε, το Συμβούλιο ήθελε μόνο του να το προχωρήσει. Όμως θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ότι δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε σε λιγότερο από 100 μέρες ε, από τις, ε, την ημέρα της οικονομικής μας υποχρέωσης ήδη θα πρέπει άμεσα το Δεκέμβριο να πληρωθούν μισθοί. Όταν λοιπόν κάνουμε ε, όταν μιλάμε για ερευνητικού οργανισμούς και τέτοιου είδους έργα, οι 100 μέρες δεν είναι τίποτα. Ε, πόσο μάλλον που έχουμε και παράλληλη συζήτηση και για το ε, πρόγραμμα ατομική ενέργειας. Είναι πάρα πολύ ε, σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα και αυτό δεν είναι καλό. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βρεθούν τα χρήματα, αλλά όχι σε βάρος του SP7. Η απόφαση για το ίτερ θα πρέπει άλλωστε να επηρεάσει και το ε, έβδομο πρόγραμμα γιατί και από το ε, ΙΤΕΡ λαμβάνονται ε, χρήματα και θα λείψουν την 1η Ιανουαρίου χρήματα. Θέλω να συμφωνήσω με την εισηγήτρια και νομίζω ότι αυτό είναι ένα, καλό, ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Η Αγγέλικα Νίμπλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη παρατήρηση, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ε, συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια. Δεύτερον, οι συνάδελφοι είπαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό να συνεχιστεί ε, στην Ευρώπη, να το διατηρήσουμε, να δείξουμε ότι και οι Ευρωπαίοι μπορούν ε, να ε, προχωρήσουν επιτυχώς σε ένα μεγάλο έργο όπως το ΙΤΕΡ και τρίτον, που είναι πολύ σημαντικό και στη γνωμοδότηση και αναφέρεται στο σημείο 4, το έργο ήταν να χρηματοδοτηθεί από το περιθώριο που απομένει. Ε, να μην γίνουν δηλαδή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα αλλαγέ. γιατί χρειάζεται και αυτό όπως και άλλα ερευνητικά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τη γνωμοδότηση συμφωνώ με την εισηγήτρια ειδικότερα σε δύο σημεία. Ε, το διωγγούμενο κόστος του ΙΤΕΡ μας απασχολεί όλους πάρα πολύ και συμφωνώ και με άλλους συναδέλφους που είπαν ότι δεν πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε από το FP7. Θα πρέπει το πρόγραμμα, δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε στρατηγικές σκέψεις για τη μείωση του κόστους. Και χαιρετίζω τα σχόλια της κυρίας Καρβάλιο και της ε, κυρίας Χέρτσογκ σχετικά με τη χρήση του προγράμματος JET. Μπορούμε να περικόψουμε δαπάνες συνολικά για το ITER αν αφήσουμε το έργο JET να συνεχιστεί και κάνοντας τις ε, προπαρασκευαστικές ε, ε, τεχνικές, νέες τεχνικές. Αυτό νομίζω ότι θα περικόψει οι δαπάνες για το ίτερ μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε. να μην υπονομεύσουμε τη χρηματοδότηση του τζέτ, γιατί θα δημιουργηθεί πολύ δυσάρεστη κατάσταση ενώ ο κόσμος εκεί που εργάζεται Είναι μακροπρόθεσμο το, έργο αυτό. Για να απαντήσω στον κύριο Όντι, να τονίσω ότι η σύνδεξη είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι εις ό,τι αφορά τους δύο βαθμούς Κελσίου για την αλλαγή στο κλίμα σε σχέση με το 2020 και οι, αλλαγές, και οι επιστήμονες ε, στο JET και στο ITER δεν πιστεύουν ότι μέχρι το 2040 θα υπάρξει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό μιλάμε για το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των έργων αυτών. Ο κύριος Σέλλαρ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, προειδοποιώ να μην πειράξουμε τα νούμερα στο ίτερ. Είναι ρεαλιστικά στην έδρασή τους, χωρίς μεγάλα αποθεματικά όμως. Και οι ισχυρισμοί ότι μπορούμε να ε, κάνουμε περικοπή για λόγους ε, δημοσιονομικούς δεν είναι σοβαρή πρόταση θα πρέπει να βρούμε ενδεχομένως μια συμβιβαστική λύση. Αλλά δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι το ίτερ θα γίνει φτηνότερο έργο αν κάνουμε το α και το β. Αυτά τα κονδυλία τα χρειαζόμαστε αυτά που έχουν αποφασιστεί. Γιατί τώρα είναι ρεαλιστική η βάση του έργου. Δεύτερον, όλα αυτά ήταν προβλέψιμα. Στις τελευταίες συζητήσεις το Κοινοβούλιο είπε για το FP7 ότι ε, αυτά τα έργα που περνάνε από την φάση της έρευνας στη φάση της ε, εγκατάστασης ε, δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από το τρέχον ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν όμως ε, πολέμησαν τη θέση αυτή του Κοινοβουλίου και είπαν ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρουμε. Ήδη πέρσι είχαμε καταλήξει στη συμβιβαστική λύση σε αυτό το θέμα και οι φιλελεύθεροι το τορπίλησαν. Το ήταν ε, ε, δεν επιλύθηκε, ενώ από πέρσι θα μπορούσαμε να είχαμε βρει μια λύση. Τα έχουμε το Ήτερ, το Γαλιλαίο, το GMS, e μεγάλα ερευνητικά έργα που περνούν στη φάση της εγκατάστασης όμως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε από το τρέχον ε, πρόγραμμα για την έρευνα. Χρειάζεται ιδιαίτερη ε, γραμμή του προϋπολογισμού ε, για τα έργα ε, για την Ευρώπη 2020. Αλλιώς το πρόβλημα θα το έχουμε και με άλλα έργα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σύντομα η Κομισιόν, σύντομη απάντηση, κυρίως να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έγιναν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για ένα άρτιο κείμενο σωστά συνταγμένο, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στην ανάγκη επίτευξη συμφωνίας για την επιπλέον χρηματοδότηση σύντομα. Τι θα πει σύντομα όμως, σε ό,τι αφορά το τζετ, αρχές του επόμενου χρόνου θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταβάλουμε μισθούς. Χρειάζεται όμως να επιτευχθεί νωρίτερα συμφωνία ή δυνατόν. Θέλω να υπογραμμίσω το ότι μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα υπάρχει το Συμβούλιο του ΙΤΕΡ και η θέση της Κομισιόν εκεί θα μπορούσε να αποδυναμωθεί λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για την πρόσθετη χρηματοδότηση. Άρα θα μπορούσαν να μας θεωρήσουν αναξιόπιστους εταίρους σε σχέση με άλλους εταίρους εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Από αυτήν την έννοια θα θέλαμε να έχουμε συμφωνία, την εντολή δηλαδή, για να διαπραγματευτούμε στις 19 Οκτωβρίου στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου. Και έχουμε και την σχετική εντολή από την Επιτροπή Κόμπου. Τώρα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και στα δύο επίπεδα, και στο διεθνές επίπεδο, στο επίπεδο του ίτερ δηλαδή, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως έχει ήδη φανεί ε, στην έκθεση πρόοδου για το έργο Fusion for Energy, έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδες στον τομέα της διαχείρισης, της εξοικονόμησης ε, και συγκράτησης του κόστους και θα το εκθέσουμε αυτό και στο Συμβούλιο. Αυτό που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι ο Διευθυντής του Fusion for Energy να έρθει στο Κοινοβούλιο και να εκθέσει τις προόδους που επιτελέστηκαν στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρατήρηση για τον σεισμό στην Ιαπωνία που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ε, και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συμβολή. Η δική μα θέση είναι ότι δεν υπάρχει άμεσο συσχετισμό μεταξύ μια φυσική καταστροφή στην Ιαπωνία ή στην Ιαπωνία και τη ε, συμβολή τη Ευρατόμ σε αυτό το έργο. Κατά συνέπεια, δεν βλέπει ανάγκη η Κομισιόν να αλλάξει ο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος Fusion for Energy για τα επόμενα χρόνια. Άρα πετούνται πρόσθετα κονδύλια, Όπω σα ε, επισήμανα και νωρίτερα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που επισπεύδω τις διαδικασίες. Ε, λοιπόν, 18 ε, Οκτωβρίου ε, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Λάβετε το υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης, μια σύντομη ανακοίνωση για να ξέρετε όλοι. Ε, Υπάρχει ένα email από συναδέλφου που παραπονούνται ότι δεν άλλαξα τη μερίσια διάταξη. Κυρίες και κύριοι, για να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ τηρώ τους κοινοβουλευτικούς κανόνες ε, και τη διαδικασία στην αρχή της συνεδρία σω δεν είσαστε όλοι εδώ. Δεν φταίω εγώ αν καθυστερήσατε να έρθετε. Ρώτησα, υπήρχαν αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Δεν υπήρχαν. Ε, αποφασίσαμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και ε, νομίζω ότι δουλέψαμε σωστά από κοινοβουλευτική και δημοκρατική άποψη. Παρακαλώ πολύ... Ε, μην ε, προβαίνετε σε τέτοια μέτρα. Ε, πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ το πρόβλημα αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να επεξεργαστούμε την ημερήσια διάταξη με τρόπο ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται δίκαια και τις και οι μεγάλες και οι μικρές ομάδες. Προσπαθώ να τις αντιμετωπίζω ισότιμα και αν δεν συμφωνούν οι ομάδες ε, μπορούμε να συζητήσουμε λεπτομέρειες. Αυτή η μέθοδος όμως παρέμβασης ε, δεν μου αρέσει. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Περνάμε στο επόμενο θέμα, ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Αλλά δεν χρειάζεται. Υπερασπίζομαι μόνος μου τον εαυτό μου. Ο κύριος Μετσάρος, εισηγητής, έχει το λόγο μόνος. Ευχαριστώ θα πρότεινα να δούμε τα δύο σημεία, το 5 και το... Συγγνώμη, το 6 και το 7 από κοινού, Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δηλαδή, να δούμε τα δύο σημεία σε ένα. Θα πρότεινα, αν δεν σας πειράζει. Για να γλιτώσουμε χρόνο. Λοιπόν, ε, σε σχέση με το με την νέα καθεστώ ε, προστασία ευρεσιτεχνιών. Συμφωνώ με του συναδέλφου που λένε ότι βιώνουμε ιστορική στιγμή τώρα. Από το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε χωρί επιτυχία να εθιτήσει ένα νέο σύστημα για διπλώματα ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας της αληθινής ευρωπαϊκής πατέντας και καλωσορίζει την πρόταση της Κομισιόν που προσφέρει μια ισορροπημένη και εφικτή λύση. Να δούμε τι νομοθετικά βήματα έγιναν στο παρελθόν λόγω δυσκολιών στο να καταλήξουμε σε ομόφωνη συμφωνία στο Συμβούλιο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις και πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις διευθυντήσεις με συγχωρείτε, οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν. 12 κράτη-μέλη ζήτησαν από την Κομισιόν να υποβάλει μία πρόταση για να εγκρίνει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα ε, του ενίου κοδεστώτο προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Ε, ε, η Κομισιόν παρουσίασε ένα πακέτο δύο νομοθετικών προτάσεων που θα επιτρέψουν σε οποιοδήποτε εταιρεία ή άτομο ε, να προστατεύσει τις εφευρέσεις του μέσω ενέως ενέου καθεστώντος προστασία φιλιστοχνιών που θα ε, ισχύει στην επικράτεια 25 κρατών μελών. Μετά από συζητήσεις, ε, τα κράτη-μέλη εκτός από την Ιταλία και την Ισπανία κατέληξαν σε μια κοινή θέση ότι για την ολοκλήρωση της ε, ε, εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητο το νέο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνίων. Το νέο καθεστώς ε, θα συνεπάρχει με τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνία που δίνονται από τα γραφεία των κρατών μελών και με το ευρωπαϊκό δίπλωμα που θα δίνεται από την σύμβαση του ευρωπαϊκού διπλώματος Ευρεσιτεχνία. Τα κράτη-μέλη και με τα ευρωπαϊκά όργανα θέλουν να δημιουργήσουν ένα ενίο πλαίσιο για το ενίο καθεστώς προστασίας ευρεσιτεχνιών για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή καινοτομία, η δημιουργία ενός τέτοιου νέου καθεστώτος ε, καταρχήν θα επιφέρει απλούστευση του σημερινού τόσο που τη χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Αυτό θα επιτρέψει στους χρήστες ε, να περικόψει το διοικητικό άχθος, θα μειωθεί το κόστος των ευρυστεχνιών ε, στην Ευρώπη μέχρι 80%. Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία που επιτεύχθη μέχρι το σαντί θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αμελητή ε, μόνο με κάποιες μη ουσιαστικές αλλαγές που μπορεί να βελτιώσουν περαιτέρω την πρόταση. Όπως ε, ως Επιτροπή εμείς για τη βιομηχανία και την ενέργεια θα πρέπει καταρχήν να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες για τη βιομηχανία και επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν ζητούν έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας γιατί θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό αριθμό των πρωταγωνιστών στην αγορά πρέπει να υπερβούν πάρα πολλά διοικητικά και οικονομικά εμπόδια. Συμφωνώ με την πολιτική της ε, κατανομής ε, των τελών ανανέωσης μεταξύ κρατών μελών και του ΕΠΟ ε, με έναν ισορροπημένο τρόπο. Αυτό είναι υπό εξέταση. Σήμερα το συνολικό κόστος της επικύρωσης για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα τεχνίας εκτιμάται μεταξύ του 22 και 26.000 ευρώ η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πατέντας ενό ευρωπαϊκού διχρώματος τεχνίας θα βοηθήσει να μειωθεί το κόστος αυτό ε, στα 680 ευρώ ανά δίπλωμα ευρεσιτεχνία και θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ε, για ε, τις επενδύσεις και την έρευνα και την ανάπτυξη. Και τέλος πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο ως ε, συνομοθέτης ε, πρέπει να τηρείται δεόντως ενήμερο για οποιαδήποτε πτυχή των υποχρεώσεων της Κομισιόν ε, προς τους νομοθέτες, τους υπόλοιπους νομοθέτες για τον κανονισμό αυτό. Τώρα θα περάσω στο δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές σχετικά με διπλώματα βρισιτεχνίας σε σημείο αυτά και θα κάνω κάποια σχόλια για αυτό το ενοποιημένο σύστημα. Ε, για να ενδυναμώσουμε την ασφάλεια δικαίου στον τομέα της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η δημιουργία ενός ενίου συστήματος επίλυσης διαφορών ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ως ε, συντάκτης της Επιτροπή ΣΥΤΡΕ προσπάθησα να παρουσιάσω κάποια στοιχεία που αφαιρούν ε, το μελλοντικό δικαιοδοτικό σύστημα ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Θα πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου και τα τέλη ε, να είναι λογικά. Ε, εμείς καλωσορίζουμε την προσέγγιση της συμφωνίας ε, γιατί βοηθά τα μέρη να ε, ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω μιας ένομης διαδικασίας. Ε, στον ενδιαφερόμενο κράτη μέλους. Επίσης, θα μπορούν ε, οι δικαστές, θα πρέπει οι δικαστές ε, να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και να λαμβάνουν συνεχή κατάρτιση. Υπάρχει ανάγκη για προτιμησιακή μεταχείριση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων υπό τη μορφή ενός μιας πιο απλοποιημένης δομής ε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη συνθήκη χωρίς χρονοτριβή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφο Γκύρακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξο όσο ο συνάδελφος ε, Μεσάρος, ε, διότι Ουσιαστικά με τον κανονισμό αυτό δεν θα πετύχουμε αυτό το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία για το οποίο αγωνιστήκαμε πριν από κάποια χρόνια. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και αυτό πραγματικά είναι μια κακή είδηση για τι οικονομίε μα. Χρειαζόμαστε επίση καινοτόμε ε, καινοτόμα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Δεν μιλάω μόνο για τα νομικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε και καινοτόμε μορφέ. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, αλλά κάποιες, κάποια ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνία στον τομέα των φαρμάκων παραδείγματος χάρη έχουν 800 ε, σελίδες. Είναι απαράδεκτο αυτό και καταλαβαίνετε και ότι επιβαρύνει σημαντικά και τη μετάφραση, το κόστος μετάφρασης. Πώς να βελτιώσουμε τους δείκτες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε και το μεταφραστικό κόστος. Αυτό που κάνουμε σήμερα βέβαια είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Απολουστεύουμε τις ταπανηρές διαδικασίες και μειώνουμε ελαφρώς το κόστος, το οποίο βαρύνει ένα μη ενωσιακό φορέα, το τονίζω αυτό, που είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρυσιτεχνίας. Επομένως, ε, μειώνουμε λίγο το κόστος, ε, το κόστος για την ε, απόδειξη του νοτερισμού, του νοτερικού χαρακτήρα μιας εφεύρησης κτλ. Πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Αυτό το ενίο καθεστώς δεν είναι προσβάσιμο ακόμη για τις ΜΜΕ και έτσι οι τρίτε χώρε, ε, οι επιχειρηματίε τρίτων χωρών θα εκμεταλλευτούν αυτό το θέμα και μπορούν να αγοράσουν άδειε στην Κίνα ή στη Ρωσία. Ο κανονισμός λοιπόν θα ήταν ε, λογικό, θα είχε νόημα αν συνοδεύεται και με την εναρμόνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σε όλες τις χώρες οι οποίες διέπονται από αυτό το ενίο καθεστώ προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Κάποιε φορέ ξέρω ότι υπάρχουν παρεκκλήσεις από την σύμβαση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δεν είναι φιλόδοξο αυτό. Βέβαια, εμείς μπορούμε μόνο να γνωμοδοτήσουμε και να εξετάσουμε τις επιπτώσεις για έναν, επαναλαμβάνω, μη ενωσιακό φορέα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Έρχομαι στο δεύτερο έγγραφο, το οποίο αφορά το δικαιοδοτικό σύστημα. Και εδώ δεν έχουν οριμάσει τα πράγματα, ούτε υπήρξε συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου έκπληξη. Αυτό το οποίο προσπαθεί εδώ ο εισηγητή να προωθήσει είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν γίνεται καθολικά αποδεκτό. Ούτε καν μεταφράσεις υπάρχουν. Η νομική γλώσσα είναι δύσκολη, είναι πολύπλοκη. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να βιαστούμε Ουσιαστικά γίνεται μια απόπειρα να γίνει κάτι επιζήμιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν έχουμε καμία αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων, των επιπτώσεων στις οικονομίες των χωρών μας. Επιχειρείται λοιπόν εδώ το κόστος ενός μη ε, ευρωπαϊκού οργανισμού που έχει δαπανηρή δράση να μεταφερθεί, να μετακυλιστεί σε βάρος τελικά των Ευρωπαϊκών φορολογουμένων. 10.000 ευρώ είναι ο μηνιαίος κατά μέσο όρο μισθός των υπαλλήλων του γραφείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένα στρατό ανθρώπων που ελέγχουν τα πράγματα, που κοιτούν νούμερα, στοιχεία κτλ. Ευχαριστώ κύριε Σφερνόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το κείμενο το ερμηνεύω ως προσπάθεια επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του κυρίου Μετσάρος σε αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά που συζητάμε για το θέμα αυτό και ε, ειλικρινά πρέπει να πούμε ότι αυτή θα είναι μια μακρά διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με όλα του τα συμπαρομαρτούντα. το οποίο θα παρέχει επαρκή προστασία σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Είναι περίπλοκο το θέμα. Βλέπουμε πόσο χρόνο τώρα συζητούν τα κράτη-μέλη. Αυτό αποδεικνύει την περιπλοκότητα της διαδικασίας που θα κρατήσει ακόμη πολύ. Η έκθεση κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μια ερώτηση ή σχόλιο σύντομο. Κατανοώ τις προσπάθειες του κυρίου Μεζάρος για, για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πράγματι, τα κόστη εδώ πρέπει να είναι λιγότερα για να μπορούμε να διαθέσουμε τους σπόρους ε, και ανθρώπινους για την ευρωπαϊκή πατέντα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να το δούμε καλύτερα το θέμα του μικρότερου κόστους για τις ΜΜΕ. Πάντοτε όταν αξιολογούμε τις ΜΜΕ κάνουμε προσπάθεια να τηρούμε κάποια όρια. Αλλά είναι δύσκολο να ελέγχουμε αν πρόκειται, για παράδειγμα, για μικρή ή μεσαία επιχείρηση κάθε φορά. Και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών θα πρέπει να προσπαθεί πάντα να βρίσκει μια ενδιάμεση λύση. Χαίρομαι διότι ο κύριος Μεσάρος μιλάει για τις ΜΜΕ εδώ γιατί αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν προβλήματα. Ίσως όμως την υποστήριξη των ΜΜΕ μπορούμε να την δούμε διαφορετικά. Είμαι βέβαιος άλλωστε ότι δεν θα είναι αυτή η τελευταία έκθεση για αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε πολλά θέματα ακόμη και πολλές εκθέσεις μέχρι ότου επιτύχουμε την προστασία της διανοητικής ε, ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Όπως σας είπα, εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του κυρίου Μεσάρος που ε, επιχειρεί να κάνει ένα βήμα ακόμη ε, στην δύσκολη αυτή πορεία προς την προστασία διπλωμάτων ευρωεσιτεχνίας. Ευχαριστώ και χαίρομαι που συνεχίζεται η συζήτηση αυτή και αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε έναν ορθολογικό δρόμο που θα λύνει ε, το πρόβλημα της ευρωπαϊκής προστασίας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά παρακαλώ όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίρεκ έχει δίκιο. Βέβαια τώρα δεν θα πρέπει να επαναλάβω κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γκίρεκ σε μεγάλο βαθμό. Όμως, ίσως ε, το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ και χρόνια περιμέναμε κάποιο αποτέλεσμα και στο πλαίσιο της Επιτροπής Ήτρε. Δεν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε και ε, αν δεν γίνουν ε, σεβαστά όλα αυτά τα κριτήρια. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εισηγητή μας. Πρέπει πλέον να βρομολογηθεί αυτό. Περιμένουμε χρόνια τώρα. Υπάρχουν κενά. Πρέπει να τα αναφέρουμε, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα την τελεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να εκκινήσουμε. Ευχαριστώ. Περιμένουμε αυτή την πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περίπου εδώ και δέκα χρόνια προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο καθεστώς ε, προστασίας των πιστοτεχνιών. Ε, και μέχρι τώρα δεν καρποφόρησαν οι προσπαθίες μας ε, και από ό,τι φαίνεται ότι τώρα έχουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Φυσικά από την αρχή είναι αδύνατο το σύστημα που θα δημιουργήσουμε να είναι τέλειο, αλλά πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εγώ γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι όταν ε, συναντώ εκπροσώπους του εμπορίου και της βιομηχανίας. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, επαρκή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και πιστεύω ότι η πρόταση αυτή έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξοδεύει κάποια ξοδεύει ε, εκατομμύρια αφενός ε, σε ε, σχέδια έρευνας και από την άλλη υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ελπίζω να επιδείξουν τα αρμόδια όργανα την απαραίτητη πολιτική βούληση για να προθεθεί αυτό το έργο. Βιντάλ Κουάντρας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το μέσο ανταγωνιστικότητας είναι απολύτως απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ενιαίο καθεστώς ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επιφέρει διάφορα πλεονεκτήματα ως προς την ανταγωνιστικότητα. έτσι ώστε και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να προστατεύσουν τα προϊόντα τους για την πνευματική τους ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπως ε, και επιχειρήσεις που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από το εξωτερικό και θέλουν στην δική μας επικράτεια να προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία για αυτές τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητο αυτό το μέσο. Κάθε φορά μιλάμε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Κάθε φορά που μιλάμε για τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε αναφέρεται η αναγκαιότητα ενό ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματο ευρεσιτεχνία. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι κανεί το αμφισβητεί αυτό. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Με την αφετηρία αυτή, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αυτό το κοινό στόχο με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη γλωσσική ετερογένεια και υπάρχει και μεγάλη ετερογένεια ως ε, προς ε, την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ε, υπάρχουν χώρες που χορηγούν πάρα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ άλλα κράτη-μέλη χορηγούν λιγότερα. το ότι δεν ε, μπορούσε να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία μας ε, οδήγησε σε, μια σε ένα απελπισμένο ελιγμό να ακολουθηθεί η ενισχυμένη συνεργασία. Όμως ε, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτελέσουμε αυτό το έργο γιατί από τις συνθήκες προκύπτει με σαφήνεια ότι το κλωσικό καθεστώς θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίζεται. Πέραν αυτού, το σύστημα της επίλυσης διαφορών ήδη έχει αμφισβητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι να προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία τη ενισχυμένης συνεργασίας κατά της οποίας ε, προσέφυγε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κάποιο κράτος μέλος, ε, δεν νομίζω ότι είναι μια παραγωγική οδός. Εγώ, Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα έπρεπε με ένα δημιουργικό τρόπο να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μία διέξοδο. Μία λύση που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή για όλους. Και ε, θα προτείνω εγώ εδώ ότι ίσως η διαδικασία των τριών γλωσσών που προωθείται τώρα μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας θα μπορούσε να ειδωθεί ως μια προσωρινή απόδειξη με έναν ορίζοντα που θα έχουν όλοι δεκτεί, δηλαδή να θέσουμε κάποια χρόνια ως ορίζοντα για να έχουμε τελικά μόνο αγγλικά. Νομίζω ότι αν όλοι το δέχονταν αυτό, τότε το τρίγλωσσο σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στάδιο μεταβατικό εισαγωγής ε, έτσι ώστε μετά από ένα λογικό χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε μία γλώσσα μόνο. Σε ένα σύστημα με μία γλώσσα μόνο αγγλικά και έτσι ώστε όλοι να είναι ισότιμοι. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή να είναι μία συμβιβαστική λύση για να βρούμε μία διέξοδο. Αν ε, επιμένουμε όλοι στη δική μας γλώσσα και δεν ε, δεχτούμε το τρίγλωσσο αυτό σύστημα και προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στη συνέχεια παραλύσουμε την όλη διαδικασία και από την άλλη πλευρά οι υπόλοιποι επιμένουν στο να διατηρηθεί το τρίγλωσσο σύστημα, δεν ε, θα είμαστε καθόλου παραγωγικοί. Εγώ προτείνω λοιπόν αυτή την οδό. Το τρίγλωσσο σύστημα να είναι ένα μεταβατικό στάδιο, εισαγωγικό στάδιο, για να καταλήξουμε τελικά μόνο στα αγγλικά. Καρβάλιο. Κύριε Καρβάλιο. Thank you very much. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε τη ρυθμίση αυτή, τον κανονισμό αυτό και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτέχνης για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εμείς ως Πρωτογαλία έχουμε προσχωρήσει στην ενισχυμένη συνεργασία. Θα προτιμούσαμε ωστόσο το γλωσσικό καθεστώς ε, να είναι μόνο αγγλικά. Και στηρίζουμε και την ιδέα του ότι θα μπορούσε το τρίγλωσσο σύστημα να είναι μεταβατική φάση μέχρι ότου περάσουμε μόνο στα αγγλικά. Έτσι θα είμαστε όλοι ε, σε ισότιμο επίπεδο, εκτός βέβαια του Νομένου Βασιλείου που ως συνήθως ε, είναι σε, σε καλύτερη θέση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σε κοινοποιήσω γιατί δεν επιθυμώ πλέον το λόγο, γιατί οι συνάδελφοι είπαν ακριβώς όσα ήθελα να πω. Έτσι λοιπόν εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βιδαλκό Άνδρες και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μπορούμε να ε, κλείσουμε αυτό το σημείο στη μερίσια διάταξη ή επιθυμεί άλλο το λόγο. Ο κύριος Μετζάρος. Ναι, να ευχαριστήσω μόνο όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τα επικριτικά και τα υποστηρικτικά. Σκοπό Ευθύμως δεν έθεσα το γλωσσικό πρόβλημα που είναι πολύ λεπτό θέμα. Είδα ότι πολλές διαπραγματεύσεις απέτυχαν ε, λόγω του γλωσσικού. Συμφωνώ όμως με την ε, διαδικασία σε μια γλώσσα στο μέλλον. Τώρα πώς θα φτάσουμε εκεί δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Ε, να πω ότι η προθεσμία είναι η 11η Οκτωβρίου για την κατάθεση τροπολογιών και για τις δύο οπότε προσανατολιστείτε ανάλογα. Πάμε στο σημείο 8, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στον Τέρμπαν. Ε, αναφερθήκαμε σε αυτό και γραπτός μεταξύ εισηγητού και σκιωδών εισηγητών έγινε η προσπάθεια να υπάρξει συνένεση ο, ο κύριος Ρόμαν Σίσλι κανονικά έπρεπε να λάβει το λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός αιθούσης. Η κυρία Ρωμάνα Τσίσλι δεν είναι εδώ. Οι ισχυώδεις λοιπόν να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Σιμάνσκι πρώτος. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έρχεται η κυρία Τσίσλι. Ε, Ρωμάνα, Ρωμάνα έχεις το λόγο, η σειρά σου είναι. Ευχαριστώ πολύ συζητούσαμε το θέμα αυτό που αφορά την αλλαγή του κλίματος. Θα μιλήσω στα σλοβενικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί ψήφισμα και φέτος για να παρουσιαστεί η άποψή μας για τις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος στον Τέρμπαν. Η Επιτροπή έχει τις ίδιες αρμοδιότητες όπως και πέρσι. Έχουμε ετοιμάσει γνωμοδότηση της Επιτροπής με τη μορφή πρόσθετων τροπολογιών και ελπίζομαι να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ο στόχος ήταν από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, να υποστηριχθεί το κείμενο που επεξεργαστήκαμε και το καταφέραμε αυτό. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδες για την συνεργασία τους, γιατί τώρα έχουμε ένα αποτέλεσμα που θεωρώ ότι είναι καλό. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας ε, τηρήθησαν, ε, περιοριστήκαμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, ε, δεν προσθέτω με κάτι άλλο. Δύο καινούργια κεφάλαια προτείνουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ένα κεφάλαιο πρώτον για τη βιομηχανία και την διατηρήσιμη οικονομία και ένα δεύτερο κεφάλαιο που αφορά την τεχνολογία και την έρευνα. Προτείνουμε όμως επίσης και ορισμένες ε, διευκρινήσεις και προσθήκες σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση η οποία είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων μας. Εδώ η γνωμοδότησή μας είναι ότι η αλλαγή του κλίματος δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως απειλή αλλά και ως ευκαιρία. Βεβαίως θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι κάνουν οι τρίτες χώρες, διότι όταν παίρνουμε μέτρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για την αλλαγή του κλίματος, τότε μπορεί να κάνουμε λάθος σε διεθνές επίπεδο και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες με τη σειρά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζουμε λοιπόν την ανάγκη λήψης μέτρων σε διεθνές σε διεθνές επίπεδο. Ε, μιλάμε επίσης για την διαφυγή άνθρακα, εκφράζουμε ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις ενεργειο, τους ενεργειοβόρους κλάδους, τονίζουμε το ρόλο της Κίνας και τον ΙΠΑ ε, σε αυτό το τομέα. Και αυτή τη φορά ε, προτείνουμε μια τομεακή προσέγγιση και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται αυτό στον Οδικό Χάρτη 2020. Μιλάμε επίσης και για την διεθνοποίηση των μηχανισμών της αγοράς. Είμαστε πεπισμένοι ότι τα κράτη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μηχανισμούς αγοράς για τη μείωση των εκπομπών και θα πρέπει να έχουν και διεθνή διασύνδεση τα μέτρα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τάχθηκε υπέρ του συστήματος ETS, εμπορίας ε, ε, εκπομπών. Στην ενέργεια και την έρευνα τονίζουμε την ε, εφαρμογή μεταφοράς τεχνολογίας με αντίστοιχη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γνωρίζουμε ότι στο Κανκούν εγκρίθηκε ένας μηχανισμός τεχνολογίας και θέλουμε να προχωρήσει στην εφαρμογή του και το ταχύτερο δυνατόν και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει ε, να επενδύονται κονδύλια στην έρευνα και την ανάπτυξη γιατί θα, πετύχουμε μόνο αν καταφέρουμε να επιτελέσουμε πρόοδο στις τεχνολογίες. Και βεβαίως ε, η μεταφορά τεχνολογίας και η μεταφορά της τεχνογνωσίας και οι αντίστοιχες επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές. Αυτά για το περιεχόμενο. Όμως κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω και δύο διαδικαστικές παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το ρόλο της Επιτροπής Ήτρε κατά την έγκριση του ψηφίσματος πριν από το Δεκέμβριο. Το για το ψήφισμα αυτό είναι αρμόδια η Επιτροπή Ένβη. Εμείς ετοιμάζομαι διευκρινιστικές ε, τροπολογίες και ο ρόλος μας ε, δεν είναι ισότιμος με εκείνον της ΕΝΒΗ. Πρέπει όμως να είμαστε ισότιμοι. Η ΕΝΒΗ καλύπτει περιβαλλοντικά θέματα. Εμείς καλύπτουμε θέματα τεχνολογικά, ενέργειας, βιομηχανίας, έρευνας, ε, τεχνολογία της πληροφορίας, όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά. Θα, τουλάχιστον το ίδιο σημαντικά όπως και τα οικολογικά θέματα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ισότιμο ρόλο Πρέπει να γίνει αυτό επισήμως, αν όχι φέτος, οπωσδήποτε του χρόνου. Και ως συντάκτρια ε, της, ε, του ψηφίσματος ε, θα πρέπει να αναδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο οι δύο επιτροπές ΕΝΒΙ και Τώρα για για την, στην Επιτροπή αλλά για την αλλαγή του κλίματος. Πόσοι είναι στην αντιπροσωπεία. Ε, ορισμένοι έχουν διαπιστευτεί. Ε, συνήθως από την Κομισιόν γινόταν αυτό μέχρι τώρα, αλλά κάθε χρόνο αυξάνονται οι δυσκολίες και το φέτος υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες από πέρσι και φαίνεται ότι οι βουλευτές που δεν είναι στην επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου μέσω της, δεν μπορούν να διαπιστευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό συνιστά πρόβλημα μεγάλο, διότι οι επιτροπές Ήτρα και ΕΝΒΗ δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η ΕΝΒΗ έχει περισσότερες έδρες στην αντιπροσωπεία από ό,τι η Επιτροπή Ήτρε. Και εκείνοι που ε, αφιέρωσαν τόσο χρόνο σε αυτά τα θέματα από την Επιτροπή αυτή δεν έχουν επίσημη διαπίστευση. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα αρνητικό είναι ότι μας δόθηκε η σύσταση να προσπαθήσουμε να διαπιστευτούμε μέσω του Globe. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε τη δυνατότητα αυτή και να μας βοηθήσει κάποιος στην διαδικασία της διαπίστευσης. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ερώτημα πρώτο. Εγώ ως βουλευτής, αν διαπιστευτώ μέσω του Globe τι θα κάνω στον Τέρμπαν. Θα έχω τις ίδιες δυνατότητες να δουλέψω και όπως και οι συνάδελφοί μου. Θα μπορώ να συμμετέχω σε όλες τις συνεδριάσεις που θα πηγαίνουν εκείνοι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, η ανεξαρτησία μου. Διότι αν εγώ διαπιστευτώ μέσω του Globe, τότε θα μου μείνει η ταμπέλα ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα σαφές ε, αν ε, είναι μη κυβερνητική ε, οργάνωση. Τι θα σκεφτεί κάποιος αν πάει σε, μια, σε ένα συνέδριο πληροφορίας και επικοινωνίας και διαπιστευτεί από τη Microsoft. Δεν είναι απλό. Ε, θα πρέπει να διασφαλίζεται, κύριε Πρόεδρε, ότι τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε που ασχολούνται με αυτές τις θεματικές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες εργασίας εκεί όπως και τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρω με όσα είπε η κυρία Συγήτρια, κυρίω τις τελευταίες ε, φράσεις τη. Και η Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί η κλιματική πολιτική θίγει και τη βιομηχανία. Έτσι λοιπόν οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν άμεση επίπτωση και στη βιομηχανία και οι συνέπειες αυτές είναι τεράστιες ε, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ αντιγωνιστικότητας ε, των βιομηχανιών μας ε, και κυρίως των ενεργοβόρων βιομηχανιών μας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, γι' αυτό η δική μου πολιτική ομάδα αναμένει τα θέματα αυτά να τα έχουμε συνεχώς κατά νου και υπό εξέταση γιατί οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες ε, πέρα από το θέμα της ε, μεταγκατάσταση. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων σε αυτό το τομέα και επιβραδύνεται και η καινοτομία σε αυτούς τους τομείς της βιομηχανίας. Γι' αυτό επιμένουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να εστιαζόμαστε στα θέματα αυτά. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ηγέτης ε, στους τομείς αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ναι, Entschuldigung, excuse me, I've made a Α, μισό λεπτό, πρώτα η Σκιώδης. Ε, ε κυρία Ούλτσοκ πρώτα. Ευχαριστώ. Α, πάει. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, ως ε, σκιώδης εισηγήτρια ε, από την ομάδα των Σοσιαλιστών, θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Ήμασταν ιδιαίτερα πρακτικοί στις συζητήσεις μας για την αναζήτηση μιας συμφωνίας και ήδη το πετύχαμε αυτό πέρσι. με σαφή τρόπο. Ουσιαστικά εμείς επιφέραμε εδώ ε, τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής ε, η Το ψήφισμα αυτό μιλά για την ενεργειακό τομέα και αυτή είναι η δική μας συνεισφορά. Γίνεται λόγος επίσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και σε εγχώριο επίπεδο. Εγώ νομίζω ότι όταν ε, ε, προβαίνουμε σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, ε, αυτά είναι τα δικά μας ε, πλεονεκτήματα που μπορούμε να επιφέρουμε. Και στο Κανκούν μάλιστα συζητήσαμε το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτή ήταν η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο έργο που έγινε εκεί όμως. Έχουμε και τα αποτελέσματα των εργασιών με τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ήδη κείμενα σε σχέση με την ε, αποδοτικότητα των πόρων ε, και κείμενα σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλε. Όλα αυτά εμφανίζονται σε αυτό το ψήφισμα. Επίσης, ε, αναφερόμαστε και σε μία παράγραφο στην ενεργειακή επισφάλεια, σημείο 14, σημείο 1. Και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις πολιτικές ομάδες που εργάστηκαν στο ψήφισμα αυτό. Όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι το θέμα του Green Job Leakage. Εμείς ε, είμαστε φιλόδοξοι για το θέμα αυτό, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρέπει να προσπαθούμε να βρίσκουμε αποδοτικές λύσεις όταν μιλάμε για πόρους. Όταν δεν είμαστε καινοτόμοι μπορούμε να χάσουμε θέσεις εργασίας. Και Φυσικά ξέρετε ότι έχουμε και τα αγωνιστές, ε, την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε, που επενδύουν πολλά περισσότερα στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν, δεν ε, θα πρέπει να θεωρούμε ότι επενδύσεις ε, στο περιβαλλοντικά θέματα είναι απλώς επενδύσεις κόστους, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις επενδύσεις αυτές ως και επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα από πρακτική σκοπιά δεν ε, θέτουμε ορθά σε εφαρμογή όλα αυτά τα θέματα. Εμείς ε, θεωρούμε όμως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα για τη δημιουργία μεγαλύτερων, περισσότερων θέσεων εργασίας. Όπως ε, σας είπα, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά. Τώρα, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή Βιομηχανίας, δηλαδή εμείς, να έχουμε και το δικό μας βάρος πέρα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν και η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η καθήλια αρμόδια επιτροπή. Εγώ νομίζω μέχρι τώρα τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά Πρέπει βέβαια να είμαστε σόφρονες και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία, να δούμε ποιε είναι οι δικέ μας θέσει, ποιες είναι οι αρμοδιότητε τη Επιτροπής Ήτρε και τι προτεραιότητες πρέπει να έχουμε. Πρέπει να υπάρχει όπως και να έχει συνεργασία και των δύο επιτροπών για το έργο αυτό και σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, διαπιστεύσεις. Εδώ υποστηρίζω σε υπησυγήτρια και ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα μας βοηθήσετε με κάποιο τρόπο στο θέμα αυτό. Τουλάχιστον υπάρχει ένα άτομο της Επιτροπής ε, Ήτρε που μπορεί να πράξει αυτό το καθήκον και επίση υπάρχει και ένα άτομο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, που δεν είναι διαπιστευμένο. Η Κομισιόν ε, μας είπε ότι δεν μπορούμε να μεταβούμε στη διάσκεψη αυτή πάρα πολύ, σε μεγάλο αριθμό. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ αριθμή αντιπροσωπεία. Το καταλαβαίνω αυτό, είναι λογικό, αλλά υπάρχουν μόνο δύο άτομα από δύο χώρες. Εμείς εκπροσωπούμε εδώ 27 κράτη-μέλη. Δεν είναι και τόσο μεγάλη αντιπροσωπεία. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια, δηλαδή όσοι ε, βουλευτές ε, είναι μέλη της Επιτροπής ε, Ήτρε και δεν είναι διαπιστευμένοι βουλευτές σήμερα να έλθουν εκεί ε, ως διαπιστευμένοι υπό τις με κυβερνητικέ οργανώσει. Όμω αυτό δεν είναι κάτι αποδεκτό. Θα έχουμε μια διάσκεψη που θα διαρκέσει πέντε μέρε. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάθε δυνατή λύση για να ξεύρουμε μια κάθε δυνατή συμμετοχή για να ξεύρουμε καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Thank you very much, President. I would like to... Ε, κυρία Καρβάλιο, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και τη... τους κοιόδες εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά τους. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μία πρόταση εδώ και πολύ καιρό ε, για την κεντρική προσέγγιση ε, που επιτέλους δέχθηκαν οι συνάδελφοι, πρόταση του ΕΛΚ, ότι δηλαδή αυτή η προσέγγιση, η μάλλον τομιακή προσέγγιση, sectoral approach που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να έχουμε κατά πολέμηση της αλλαγής του κλίματος αφενός μια ανταγωνιστικότητα αφετέρου και μείωση της διαφυγής άνθρακα. Και αυτό όπω είναι ένας νέος τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις και να βρούμε καινοτόμες λύσεις για μια νέα διεθνή συμφωνία η οποία θα αντικαταστήσει τη συμφωνία του Κιώτο. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω, χαίρομαι που έχουμε ένα σχεδιασμό του CDM που είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν έχει εφαρμοστεί πολύ καλά αυτός ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης και μόνο δύο χώρες ουσιαστικά έχουν επωφεληθεί, Ινδία, Κίνα. Όμως αυτός ο μηχανισμός νομίζω ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ούτω ώστε να εκπληρώσει και τη συνιστόσα την αναπτυξιακή, να βοηθήσει αναπτυσσόμενες χώρες και ίσως και παραλλήλω να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, CDM, κάνει δοκιμές κομισιών, παραδείγματο χάρη τομεακές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Κίνα ή Ινδίας. Αυτό να είναι ένα διαφορετικό σύστημα που θα λειτουργεί παράλληλα. Και τέλος, στηρίζω πλήρως αυτό που είπαν οι προλαλήσαντε συνάδελφοι για τη διαπίστευση για την αντιπροσωπεία που θα πάει στο Ντέρμπαν ο συντονιστής μας θα επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα. Ευχαριστώ. Βέρα Τελκαστήγιο, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τελευταίο σχόλιο φυσικά και προσυπογράφω τα όσα είπε η συγγήτρια και τη συγχαίρω και εγώ για το εξαιρετικό τη έργο όπως και τους κοιόδης εισηγητές. Θέλω να μείνω στα διαδικαστικά. Νομίζω ότι εδώ πολλές φορές υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το γιατί πρέπει η Ήτρε να είναι ουσιαστικά ε, παρούσα επίση ώρες με την ένβια. Έχει να κάνει με τις αλλαγές του κλίματος, αλλά υπό ένα σκέλο, υπό μία προοπτική, δηλαδή τον καθορισμό των στόχων, την καθιέρωση των προϋποθέσεων, τη θέση των προποθέσεων και των όρων ότι είναι ε, η κατάσταση που βιώνουμε έτσι όπως έχει, έχουμε την αλλαγή του κλίματος και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς ε, ως ΙΤΕΡ πρέπει να δούμε πώ μπορούν να εφαρμοστούν οι στόχοι στην πράξη. Άρα είναι αναπόφευκτο να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία των δύο επιτροπών. Βέβαια αυτό δεν ανταποκρίνεται στη σύνθεση των επιτροπών που παρίστανται σε διεθνεί αποστολέ, σε διεθνεί αντιπροσωπείε και συγκεκριμένα στις ε, διασκέψει για την αλλαγή του κλίματο. Για να είμαστε πρακτικοί, είναι λίγο ανεξήγητη κατάσταση στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ουσιαστικά τα κονδύλια ε, τα οποία έχουμε εμείς στη διάθεσή μας για να παρευρισκόμεθα σε κάποιες ε, συνεδριάσεις, ε, τελικά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάμε στον Τέρμπαν. Και υπάρχει το εξή επιχείρημα γι' αυτό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισορροπία της εθνικής εκπροσώπησης σε ό,τι αφορά τη σύνθεση ε, αναπολιτική ομάδα. Δηλαδή, Σήμερα ένας βουλευτής μπορεί να πάει να δει, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα και του λένε όχι για να πας στον τέρμαν δεν μπορείς. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Ίσως να είναι εύκολο, πολύ εύκολο. Θα μπορούσε να ληφθεί μια ισορροπημένη απόφαση για τον αριθμό των βουλευτών από κάθε ομάδα οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τους πόρους αυτούς για να μεταβούν στον Τέρμπαν. Δεν ξέρουμε σε συνάρτηση με ποιο κριτήριο για τη συγκρότηση της επίσημης αντιπροσωπείας. Τρει, δύο, ένα από την κάθε πολιτική ομάδα, δεν ξέρω και εγώ πώς. Αλλά πρέπει να έχουμε έναν ελάχιστο αριθμό μελών, μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χρηματοδοτούν μόνοι τους ε, την ε, συμμετοχή τους, αλλά η διαπίστευση είναι σημαντικό και μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική διάσκεψη. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των μελών που θα μπορούσαν να πάνε εκεί. Πρέπει να δείτε κύριε Πρόεδρε και εσείς πώς μπορούμε να το διχειριστούμε αυτό. Είναι πολύ απλό το θέμα. Πρέπει να έχουμε αντίστοιχο αριθμό βουλευτών. από την κάθε πολιτική ομάδα που απαρτίζουν αυτή την αντιπροσωπεία. Θα πρέπει να μπορούν αυτοί οι βουλευτές με χρήση δύο πόρων να παραστούν στον Τέρμπαν και να έχουν και τη διαπίστευση την απαραίτητη, να μην χρειάζεται να προσφύγουν σε άλλους οργανισμούς για να έχουν τη διαπίστευση. Είναι λίγο ανόητο, είναι λίγο γελίο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Γολάνσκα, Πουβίνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Θέλω να επαναλάβω δύο θέματα. Εγώ ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας ε, στην Ινδία και πρόσφατα επέστρεψα από μια συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι δεν αναλαμβάνουμε κανένα μεγάλο έργο με την Ινδία, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι δύσκολο να πετύχουμε μια κατανόηση σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση και ίσως κάτι τέτοιο πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε διμερή project για το κλίμα και Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και κάποιων τρίτων χωρών, όπως η Ινδία. Κάτι τέτοιο θα μας επέτρεπε να βελτιώσουμε τη δική μας προβολή και Έτσι λοιπόν δεν θα λεγόταν ότι δεν συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα μπορούσαμε να προβούμε σε κάποια ευαισθητοποίηση. Τέτοιου είδους οικονομική διπλωματία είναι πολύ σημαντική, τόσο σημαντική όσο και πολιτική διπλωματία τέτοια θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια πρέπει να βρίσκονται υψηλά στην ημερησή διάταξή μας. Πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Ένα άλλο θέμα είναι η ενισχυμένη συνεργασία. Εδώ απευθύνομαι στον Πρόεδρο. Έχω ένα αίτημα. Έχω ένα αίτημα, Πρόεδρε. Ίσως ε, ο κανόνας για την ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά. Υπάρχουν 51. Γιατί υπάρχουν ε, διάφορα θέματα που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και αφορούν και τις δύο επιτροπές μας ενίοτε. Εγώ συμμετέχω και στις εργασίες της Επιτροπής ΕΝΒΗ και μπορώ να δω η μα ότι μιλάμε για ίδια θέματα αλλά από διαφορετική σκοπιά. Αυτά τα θέματα αφορούν και τις δύο λοιπόν επιτροπές και ίσως πρέπει να χρησιμοποιούμε τον κανόνα 51 πιο συχνά. Εντάξει, θα το δώσουμε στην ΕΝΒΗ, θα το οριστικοποιήσουμε με την ψηφοφορία. Δεύτερον, συχνά, όπως είπε η κυρία Κολάσκα-Μπομπίνσκα, υπάρχει το θέμα της συμμετοχής των δύο επιτροπών σε θέματα που τους αφορούν, αφορούν και τις δύο. Συχνά συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις και έχουμε ένα σωρό διαπληκτισμούς για αρμοδιότητες, για ε, συμφωνίες, όλα αυτά ε, είναι αφόρητα και δεν οδηγούν στην επικράτηση των καλύτερων επιχειρημάτων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα δούμε καλύτερα τα θέματα αυτά, κυρίως όταν πρόκειται για τέτοια ψηφίσματα. Τα λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά, εγώ δεν ξέρω λύση ακόμα. Τέλος, το ζήτημα της αποστολής της αντιπροσωπείας ε, η διάσκεψη των Προέδρων των Ομάδων θα αποφασίσει, από εκεί θα ρυθμιστεί το θέμα γιατί υπάρχει περιορισμός. Θα ήθελα να πω ότι η αντιπροσωπεία αυτή είναι μια ειδική αντιπροσωπεία. Ε, τώρα, ε, σε άλλα θέματα το ζήτημα αυτό έχει απορριφθεί εκτός της ποσόστοσης. Άρα λοιπόν ήδη εδώ υπάρχει κάποιο προνόμιο ε, για τη διάσκεψη για το κλίμα. Υπάρχει πρόβλημα όμως για αυτούς που θέλουν να πάνε όλους μπορεί να γίνει διεπιστολών, πώς θα οριστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Μπορώ εγώ να του στείλω μια επιστολή, αλλά βέβαια το θέμα της διαπίστευσης είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και αν κατάλαβα καλά, έχει σχέση να κάνει με την αλλαγή στη στάση της Κομισιόν, γιατί παλιότερα η Κομισιόν τα έκανε όλα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν να μας εξηγήσει γιατί άλλαξε το σύστημα. Εντάξει, τώρα ξαφνικά προέκυψε το ερώτημα, αλλά ίσως μπορεί κάποιος να απαντήσει. Αν δεν απαντήσει, ίσως πρέπει να στείλουμε επιστολή στην Κομισιόν. Γιατί αυτή η διαδικαστική αλλαγή δημιούργησε τα τωρινά μας προβλήματα της διαπίστευσης. Και συμφωνώ με όλους που είπαν ότι είναι δύσκολη πρόσβαση και συνάδελφοι από το Κοινοβούλιο ε, τώρα στέλνονται να διαπιστευτούν από κάποιον άλλο οργανισμό. Αυτό δεν είναι εντάξει, δεν είναι σωστό και συμφωνώ με αυτά που είπατε. Ε, λοιπόν, εις ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχής ήτρα ένβη να στείλουμε μια επιστολή, ένα αυτό, και δεύτερον ερώτηση προς την Κομισιόν για να αριθμίσει και το θέμα της διαπίστευσης. Κυρία Ντεκαστήγιο, η Κομισιόν δίνει τη διαπίστευση μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου. Άρα το Κοινοβούλιο πρέπει να ε, πάρει την πρωτοβουλία έχοντας αποφασίσει πόσους θέλει να στείλει η Κομισιόν. Αν πούμε 100 θα πει η Κομισιόν όχι. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει το Κοινοβούλιο να διατυπώσει το αίτημα. Η διάσκεψη των Προέδρων ε, πρέπει να αποφασίσουν. Υπάρχει αυτό, το, αυτή η διαδικασία μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Εκεί πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τον αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας, όπως έχει τώρα, να είναι ο ίδιος αριθμός, η ίδια κατανομή και τα νέα μέλη της αντιπροσωπείας θα χρηματοδοτήσουν την μετάβαση από δικά τους χρήματα για να πάνε και εκείνοι στη διεθνή συνάντηση ή σε άλλες συναντήσεις. Λοιπόν, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου, σε τελευταία ανάλυση και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η διάσκεψη των προέδρων των ομάδων θα λάβουν την απόφαση. Εγώ θα παραπέμψω το ερώτημα αυτό για να το λύσουν, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο κύριος ε, Γκίρεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που μας απασχολεί. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τη λειτουργία των αγορών. Η τυποποίηση διευκολύνει τη λειτουργία των αγορών και της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και της παγκόσμιας. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στον επακριβή καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων ε, που θα πρέπει να ισχύουν στη μαζική παραγωγή, στα πρότυπα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ε, στο πλαίσιο της, ε, του ICT, των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Εδώ μιλάμε για οικονομίες κλίμακος. Αυτό διακυβεύεται εδώ. Και τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν, είναι το ερώτημα. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι να υπάρξει δέουσα αναγνώριση φυσικά και θέλουμε εναρμονισμένα πρότυπα και στις 27 χώρες μέλη. Αυτό θέλει η Επιτροπή τουλάχιστον. Θέλει να επιταχύνει ε, τη διαδικασία αυτή της καθαίρωσης των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων που είναι χρονοβόρα, δύο-τρία χρόνια διαρκεί και θέλει να καλύψει και την τεράστια αγορά υπηρεσιών αυτό το σύστημα και επίσης θέλει ε, στον τομέα του ICT επίσης να εισαγάγει πρότυπα και να δώσει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, την ε, ίδια πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση στην ανάπτυξη προτύπων και τη χρήση αυτών. Όμως ίσως αυτό αποδειχθεί και είναι άλλωστε σήμερα δύσκολο. Οι φορείς τυποποίησης, οι εθνικοί ιδίως φορείς τυποποίησης, λειτουργούν ουσιαστικά σαν φορείς της ανοιχτής αγοράς. Όμως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ουσιαστικά θα αναπτύσσονται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Φαίνεται να υπάρχει λοιπόν σύγκρουση συμφερόντων. Από τη στιγμή που η εναρμόνιση οδηγεί στη βαθμιαία κατάργηση των ε, εθνικών προτύπων προς όφελος των ευρωπαϊκών προτύπων. Και όλα αυτά με φέρνουν ε, στην εξή ερώτηση που θέλω να διατυπώσω. Η Κομισιόν θέλει τελικά να προβεί σε προοδευτική εξάλληψη των εθνικών ε, φορέων τυποποίηση Και ένα επόμενο ερώτημα. Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με τις μικρότερες πλούσιες εταιρείε σε ό,τι τα πρότυπα. Το σχέδιο κανονισμού δεν δίνει πληροφορίες τι είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο σε σχέση με ένα πρότυπο ISO, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά την παγκόσμια, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα πρότυπα επίσης βασίζονται στο copyright, στην πνευματική ιδιοκτησία. Και θα πρέπει να διατηρηθεί το copyright, αλλά μετά τη δημοσίευση μπορεί τα πρότυπα αυτά να επηρεάσουν κάποιε διαδικασίε κατοχήρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ προτύπου και διπλώματο ευρεσιτεχνία, μάλλον άδεια συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, ή τα e-standards. Τι γίνεται με αυτά. Επόμενο ερώτημα. Η, η μετάφραση κατά την εναρμόνιση των εθνικών προτύπων. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από τη, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λόγω του χρόνου και του κόστους που συνεπάγεται η μεταφρασή τους. Και επίσης πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ανάπτυξη των διαφόρων προτύπων στον τομέα των ε, τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, ε, τα διάφορα φόρα. Ε, λοιπόν, αυτά ουσιαστικά είναι τα προβλήματα τα οποία έχω εντοπίσει. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα. Η έκθεση είναι καλή, αλλά πρέπει να την επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο ακόμη. Μπαλτσίτης τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο στην Επιτροπή μας και συμφωνώ με τον συνάδελφο, με τον συγκητή, για ορισμένους ε, φόβους και μειονεκτήματα που εντόπισε Στην τρέχουσα πρόταση. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα και ανταγωνιστική αγορά, όπου κάθε παίκτη θα έχει ε, ένα σαφή ρόλο και θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνε για όλου και θέλουμε να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια, πρέπει να δημιουργήσουμε κοινέ ε, αρχέ τυποποίηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάτι τέτοιο θα μα βοηθήσει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και επίσης ε, θα μας ε, επιτρέψει ε, να αναθεωρήσουμε το όλο σύστημα δημοσίων προμηθειών, ίσως να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα δημοσίων προμηθειών δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ωφελεί όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που άκουσε τις προτάσεις μας και ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια πιο διαφανή και πιο δίκαιη ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα μπορούμε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Κύριος Βέμπερ. Και εγώ συμφωνώ με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του εισηγητή. Να προσθέσω ένα σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη νομοθετική δύναμη διαθέτει και μία αγορά 550 εκατομμυρίων αγοραστών πρόκειται για την πιο μεγάλη παγκόσμια αγορά. Έτσι λοιπόν για την πρόσβαση σε αυτή την αγορά ο σεβασμός των κανόνων που ε, θεσπίζει είναι σημαντική δύναμη το θέμα είναι ότι δεν ε, υπάρχει ε, ένας έλεγχος, δεν υπάρχει δικαστήριο που να ελέγχει. Ποιος ελέγχει ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που εκπονούμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείες το πράττουν και η Κίνα το πράττει δεν ε, διστάζουν ε, να έρθουν στις δικές μας επιχειρήσεις για να δουν πώς παρασκευάζονται, πώς κατασκευάζονται τα αγαθά και αν, γίνονται, και αν γίνεται σεβαστή η υγειονομική νομοθεσία και έχουμε μια μεγάλη αδυναμία. Το ίδιο συμβαίνει, παραδείγματο χάρη και στο τομέα τη μετανάστευση. Έχουμε νομοθεσία, αλλά δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Έτσι λοιπόν, προτείνω διαδικασίε ελέγχου και ένα δικαιοδοτικό σύστημα, έτσι ώστε να μπορούμε ε, να ελέγχουμε την εφαρμογή των όσων νομοθετούμε. Ο κύριο Σοντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατόπιν όσων ε, υποθήκαν από τον κύριο Βεμπέρ, με το οποίο συμφωνώ, Αναρωτιόμαι μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να επωφεληθούμε από αυτή την πολιτική συζήτηση για την τυποποίηση για τα πρότυπα προκειμένου να συνδέσουμε αυτό το θέμα με τη βιομηχανική πολιτική. Γιατί η εντύπωση που μπορούμε να έχουμε είναι ότι τελικά έχουμε συνεχώς κανόνες, πρότυπα ε, για τον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας ε, κτλ. αλλά δεν προσδίδουν τη ιδιαίτερη προσοχή για το ποιος ε, θα κατασκευάσει τα προϊόντα ε, που πρέπει να σέβονται αυτά τα πρότυπα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τα air condition, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάξαμε τα υγρά που χρησιμοποιούνται στα air condition. Δεν μπορώ να σας πω τώρα τίποτα παραπάνω, δεν είμαι ειδικό. Έχουμε λοιπόν το πρότυπο αλλά καθώς ε, δεν προσέξαμε ε, ποιος ε, θα τα κατασκευάσει, έχουμε εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε μία αγοραστική δύναμη που φεύγει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, γιατί η κατασκευή γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε προωθήσει με την εσωτερική μας αγορά μέσω μιας προσέγγισης τυποποίησης, όμως ε, αν θέλουμε ε, να την προωθήσουμε περαιτέρω, πρέπει να δούμε ποιο ε, θα προβεί και στην κατασκευή αυτών των προϊόντων και θα πρέπει να εφαρμόσει αυτού του κανόνε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα επαρκή έλεγχο, προκειμένου να υπάρχει πλήρη και πραγματική εκτέλεση στο σύνολο τη εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρίκμαν από την Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να πω δύο λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να πω ότι καλωσορίζουμε το σημαντικό θέμα της τυποποίησης και το, το συζητάτε στην Επιτροπή σας. Πιστεύουμε ότι μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε τα μάλλα στη συζήτηση για το πώς θα καταστήσουμε την ευρωπαϊκή τυποποίηση να λειτουργεί καλύτερα, πώς θα εξυγχρονιστεί και θα πλουστευτεί. Αυτός είναι ο στόχος της Κομισιόν και να έχουμε και το σύνδεσμο με τους διάφορους στόχους της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 σχετίζεται πολύ στενά με το δικό μας ε, στόχο να βελτιώσουμε τα πρότυπα που θα μπορούν να είναι χρήσιμα για την καινοτομία, για τη βιομηχανική πολιτική και για πολλές άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θέλουμε με το πακέτο αυτό να καταστήσουμε πιο σύγχρονο το σύστημα, να είναι πιο προσαρμόσιμο στις τεχνολογικές αλλαγές. Ε, όλες οι προτάσεις μας έχουν αυτό το στόχο. Έτσι λοιπόν, κατανοώ ότι ο εισηγητής ε, έχει κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το περιεχόμενο. Ευχαριστώ να σας διευκρινίσω ότι με τη δέσμη μέτρων ε, δεν θέλουμε να φέρουμε μια, την επανάσταση στο σύστημα τυποποίησης, θέλουμε απλώς μια εξέλιξη. Έτσι λοιπόν δεν θίγουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι εθνικοί φορείς τυποποίησης, σεβόμαστε τις κυρίες αρχές της ευρωπαϊκής τυποποίησης, δηλαδή τον εκούσιο χαρακτήρα του προτύπου, ότι πρέπει ε, να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της αγοράς ε, και ότι πρέπει να υπάρχει μία ε, ε, δουλειά τυποποίησης που βασίζεται στη δουλειά των εθνικών φορέων τυποποίησης. Αυτά τα στοιχεία δεν τα αλλάζουμε, δεν τα τροποποιούμε καθόλου. Αυτό θέλαμε να το διευκρινίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε ενδεχομένη παρεξήγηση για το τι κάνει η Κομισιόν. Δεν μιλάμε λοιπόν ε, για ριζική αλλαγή ούτε για επανάσταση. Εδώ πρόκειται για έκθεση δύο πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και προσπαθούμε εμεί να σεβαστούμε τα όσα είπε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του τον Οκτώβριο του 2010. Έτσι λοιπόν κατανοούμε το σύνδεσμο μεταξύ της τυποποίησης και της ανταγωνιστικότητας και συμφωνούμε με όσα υπόθηκαν από τους διάφορους ομιλητές για την ανάγκη να έχουμε ένα σαφή ρόλο για το ρόλο της τυποποίησης, της ασφάλειας των προϊόντων και της εποπτείας της αγοράς. Υπόθηκε ότι είναι καλό να έχουμε νομοθεσία, αλλά στη συνέχεια πώς διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα που τίθενται σε εμπορία είναι πραγματικά ασφαλή για τον καταναλωτή. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή που έμεσα σχετίζεται με την τυποποίηση, αλλά υπάρχει ένα σαφής σύνδεσμος μεταξύ όλων αυτών. Η εποπτεία της αγοράς είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Αυτές είναι υπεύθυνε για την εποπτεία της δικής τους αγοράς Υπάρχουν λοιπόν εθνικές εποπτικέ αρχές, ο ρόλος τους είναι να εξετάζουν τι συμβαίνει στην αγορά και να αποσύρουν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή ή δεν σέβονται την νομοθεσία και επίση ε, και οι τελωνίκοι στα σύνορα διαδραματίζουν ένα ρόλο. Εμείς τι θέλουμε, να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, να βελτιώσουμε την εποπτεία της αγοράς, τη σχετική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και έχουμε ήδη ένα κανονισμό για την εποπτεία τη αγορά του χρόνου. Θα παρουσιάσουμε και νέα πρόταση για να ενισχύσουμε την εποπτεία τη αγορά. Έτσι λοιπόν, για όσα υπόθηκαν, ε, τα όσα υπόθηκαν ε, σε σχέση με το σύνδεσμο εποπτείας της αγοράς και ε, βιομηχανικής πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εμεί θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιε είναι οι τομείς προτεραιότητας για την Ευρώπη όπου θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη και αυτή η δραστηριότητα περί προτύπων συνδέεται με την προτεραιότητα που δίνουμε στη βιομηχανία στο μέλλον, δηλαδή για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας μέχρι το 2020. Θέλουμε να τονίσουμε λοιπόν ότι για μας είναι σαφές ότι και η δική σας επιτροπή έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρώτη συζήτηση είναι αυτή σήμερα. Θα μην ξαναμιλήσουμε. Οπότε για τώρα κλείνουμε το σημείο αυτό και πάμε στο επόμενο που είναι το σημείο 10 όπου πρόκειται για, το θέμα προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη. Ο συνάδελφος Πατριτσέλο είναι ο εισηγητής και πρώτος θα παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής ΙΤΡΕ και συγκεκριμένα τον κύριο Μπέιερ για την διαθεσιμότητά του και την επαγγελματικότητά του, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το πρώτο στάδιο σύνταξη του κειμένου. Τώρα, το να συζητάμε την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική δύο εβδομάδες πριν από την εκτόξευση των δύο δορυφόρων του Γαλιλαίου που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου από το Κουρού νομίζω ότι μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα που συζητούμε εδώ σήμερα. Μετά από έτη προετοιμασιών ε, έχουμε την ικανοποίηση να παρακολουθήσουμε αυτό το στάδιο της εκτόψευσης. Ε, το πρώτο, η πρώτη συνιστόσα του προγράμματος που θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματική ανεξαρτησία στην δορυφορική ραδιοπλοήγηση και ε, η επίτευξη αυτού του στόχου ουσιαστικά προέρχεται και από ε, το άρθρο 189 της Συνθήκης της Λισαβόνας που με σαφή τρόπο προσδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδίδει την Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη να συντονίσει και να παγιώσει τις διαστημικές, τις εθνικές διαστημικές πολιτικές και τα εθνικά προγράμματα σε μία προσέγγιση για να ε, προωθηθεί η επιστημονική και τεχνική πρόοδος και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Ένας στόχος που τέθηκε από τη συνθήκη που αναγνωρίζει τη σημασία του διαστήματος σε κοινωνικό, οικονομικό ε, και στρατηγικό επίπεδο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει στην παγκοσμία σκηνή να μπορεί να ανταγωνιστεί με τους υπολείπους. Ε, έτσι λοιπόν η συνθήκη μας δίνει μια κατάλληλη νομική βάση ε, για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων για τους οποίους ε, τα όργανα, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταρχήν το Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους και τα κατάλληλα νομοθετήματα. Προς αυτό το σκοπό συμφωνώντας ε, με τη σημασία που έχει δώσει μέχρι τώρα η Κομισιόν στο Γαλιλαίο, έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής, ε, επιμεμβάνω ότι τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα και ο στρατηγικός ε, χαρακτήρας του προγράμματος είναι κάτι πολύ σημαντικό και από οικονομική και από στρατηγική σκοπιά. Είμαι πεπισμένος ότι μόνο μέσω μιας ε, διαστημικής πολιτικής η οποία ε, θα ε, προσδίδει αξία και στα δύο προγράμματα μπορούμε να εγγυθούμε την τεχνολογική ανεξαρτησία και την πολιτική αυτονομία της Επίρου μας ε, ε, κάτι το οποίο θα φέρει πάρα πολλά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη στους πολίτες. Ε, θα εγγυηθεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και για το λόγο αυτό εκφράζω την θλίψη μου για την απόφαση της Κομισιόν να μην ε, συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση του GMS στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ε, γνωρίζοντας ότι η έλλειψη ενός ε, τέτοιου δημοσιονομικού πλαισίου κινδυνεύει να καταστήσει άχρηστες τις επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέρα ε, από τις ε, ανησυχίες που εκφράστηκαν σε ό,τι αφορά τις ε, οικονομικές πτυχές, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την στρατηγική που θέλει να προωθήσει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις πτυχές της διαχείρισης των προγραμμάτων Γαλιλαίου και GMES προκειμένου να τα καταστήσει πλήρως επιχειρησιακά μόνο μέσω του πλήρους ακροτολογισμού ε, της οργανωτικής δομής των προγραμμάτων ε, θα μπορέσουν ε, να υπολογίσουμε το κόστος διαχείρισης και συντήρησης προσδίνοντας τους Ευρωπαίους πολίτες ένα σαφές πλαίσιο για ε, τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θέλω να τονίσω στην πρότασή μου είναι αυτό που αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ε, εποπτείας ε, του περιβάλλοντος και του διαστήματος είναι σημαντικό να εξηγήσουμε, να, συγγνώμη, να στείλουμε ευρωπαϊκούς δορυφόρους στο διάστημα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την προστασία τους ε, ε, προστατεύοντας αυτούς τους δορυφόρους από τη σύγκρουση με τους αστεροειδείς ε, και τα διαστημικά απόβλητα. Ένα άλλο θέμα ε, που πρέπει να προσέξουμε αφορά την έρευνα. Θέλουμε ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία. Θα πρέπει να επενδύσουμε και στην καινοτομία και μέσω ad hoc ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για να συντονίσει τις δραστηριότητες έρευνας των μεμονωμένων κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία προκειμένου να μην υπάρξουν επικαλύψει ε, και κενά που θα μπορούσαμε να δούμε αν δεν υπάρχει διαχείριση οργανωτική. Και ε, πεπισμένος ε, ότι ε, πρέπει να έχει ευρωπαϊκή πολιτική, αυτόνομη διαστημική πολιτική Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο η Κομισιόν ε, να καθορίσει μια στρατηγική διεθνούς συνεργασίας σε προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με ορισμένους στρατηγικούς εταίρους, Ρωσία και Ηνωμένε Πολιτείε για την υλοποίηση ε, της βιομηχανικής συνεργασίας ε, και κοινή επένδυση σε μεγάλα έργα και προγράμματα. Τέλος, θεωρώ ότι η αυξανόμενη συμμετοχή ε, της Ένωσης στο διάστημα ε, θα πρέπει να προσδιορίσει εκ νέου τις σχέσεις έχοντας κατά νου ότι οι τεχνικές αρμοδιότητες ε, και τα προγράμματα που αναπτύσσονται από τον οργανισμό είναι θεμελιώδη για τη διαχείριση της τεχνικής ικανό, τεχνολογικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή ως συντάκτης για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική. Ε, στο πρώτο αυτό στάδιο ε, θέλω μαζί και με τις δικές σας πρωτοβουλίες και με τη δική σας προσωρά να προχωρήσω ως εξή. Ε, να εκπονήσουμε μία έκθεση που θα συνάδει με το άρθρο 189 της Νέας Συνθήκης και το κείμενο αυτό να μπορέσει να εγγυάται την οικονομική και, επιστημονική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκλάντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Πατριτσέλο, για την ισορροπημένη και ωραία έκθεση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα επικεντρωθώ σε κάποια μικρά σημεία που πρέπει να ενισχυθούν ενδεχομένως ή να τα επεξεργαστούμε περισσότερο ε, δημοσιονομικά. Λοιπόν, για τη χρηματοδότηση συμφωνούμε νομίζω στο Κοινοβούλιο ότι αυτά είναι κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης. Αν θέλουμε ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική με το έγνωστο Γαλιλαίος ε, GMES κλπ. θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό ε, Προπολογισμό για να μπορούμε να ασκούμε επιρροή και να επηρεάζουμε την πορεία αυτών των έργων και προγραμμάτων. Ο παραλήπτης αυτής της συζήτησης νομίζω ότι είναι το Συμβούλιο. Βλέπω να ε, νεύει εκεί ο εκπρόσωπος της Γραμματείας του Συμβουλίου μπορούμε να διατυπώνουμε τα αιτήματά μας, θέλουμε προγράμματα ε, μεγάλης αλλά μπορεί να σκοντάψουμε στα δημοσιονομικά. Είναι δύσκολο τώρα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα με την οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά αυτά τα διαστημικά προγράμματα, η διαστημική στρατηγική δίνει προστιθέμενη αξία. Δημιουργεί θέσει εργασία, απόδοση επενδύσεων. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στα κράτη-μέλη, ότι στι δημοσιονομικέ προοπτικέ και τον προπολογισμό πρέπει να γίνουν καλοί. Ε, υπολογισμοί, γιατί οι δορυφόροι κρατάνε 5, έχουν διάρκεια ζωής 5-7 χρόνια και άμα δεν μπορούν να ε, χρησιμοποιούνται πρέπει να αντικαθίστανται. Πρέπει η καινούργια γενναία να χρησιμοποιείται και να συνοδεύονται από τις υπηρεσίες τις ε, ανάλογες. Μιλάμε για τα διαστημικά συντρίμια, επιθέσεις, μιλήσαμε για τα κυβερνοεγκλήματα, γιατί αυτά θα πρέπει να είναι δικτυωμένα, οι διορυφόροι δεν μπορεί να είναι μόνο στην ατμόσφαιρα, πρέπει να έχουν και πήγες διασυνδέσεις, είναι σημαντικό και αυτό και έχει να κάνει με επιθέσεις. Ε, από τις εμπειρίες μου, από άλλες εκθέσεις για τον Γαλιλαίο, ε, Μιλάμε για επιτήρηση συχνά και το λέει και στο σημείο 18 εδώ, έλεγχο των συνόρων, ε, επιτήρηση των συνόρων. Και εδώ δεν έχω υπόψη μου τη Frontex, έχω υπόψη μου την, πειρα, πειρατεία από την Αφρική. Εκεί πρέπει να υποστηρίζονται στρατιωτικές μονάδες με ένα ακριβές σύστημα που να μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ των αλλιευτικών σκαφών και των σκαφών των πειρατών για να καταπολεμηθεί η πειρατεία. Θα γίνουν συζητήσεις εδώ, έχουν γίνει άλλες. Το σημείο 22 είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα ε, να το στηρίξουμε ακόμα περισσότερο και μέσα από τις τροπολογίες, ε, δυνατότητες συνδυασμού, τηλεπικοινωνιακά συστήματα με δορυφόρους, Galileo, GMES, ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε καλύτερα και να αναπτύξουμε και μια στρατηγική για το συνδυασμό των υπηρεσιών ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν όλες οι υπηρεσίες. Ε, τέλος, πρέπει να το συζητήσω αυτό με τον εισηγητή, να δω τη γνώμη του. Ε, φαντάζομαι ότι θέλουμε αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Ωραία, το θέλουμε αυτό. Από την άλλη υπάρχει και διεθνή συνεργασία όμως, άρα πρέπει να σταθμίσουμε τα δύο. Δηλαδή η αυτονομία, η πρόσβαση, συστήματα εκτόξευσης και λοιπά να γίνονται, αλλά να γίνεται και η διεθνή συνεργασία και να έχουμε ανταγωνισμό. Γιατί το έχουμε ζήσει όταν ε, μειώνεται ο ανταγωνισμός ε, και αν επικεντρωνόμαστε σε ένα σύστημα ε, μπορεί οι τιμές να αυξηθούν. Αυτή την ισορροπία θα πρέπει να την δούμε. Κατά τα άλλα, συμφωνώ, είμαι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα ε, και θα πρέπει να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα συνεργάζεται με την ΕΖΑ και τα κράτη-μέλη και ΕΖΑ και κράτη-μέλη. αυτά είχα να σας πω προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρεμέκ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή διότι θεωρώ ότι έκανε πολύ και καλή δουλειά. Σε αυτά τα πλαίσια στις παρατηρήσεις μου θα επικεντρωθώ σε ορισμένες πτυχές που τις θεωρώ τις πιο σημαντικές. Πριν από λίγο κάναμε ακρόαση για το θέμα αυτό και έδειξε η ακρόαση ότι ε, όλο και δυναμώνουν οι φωνές που ζητούν πιο φιλόδοξη διαστημική πολιτική. Εμείς ε, έχουμε μια παράδοση, έχουμε μέσα, έχουμε αποτελέσματα σε αυτό το τομέα και πολύ καλούς ε, ειδικού επιστήμονες. Εκεί που δεν υπάρχει σαφήνεια είναι στις προτεραιότητες. είχαμε 50 προτεραιότητες και δυσκολευόμαστε να χρηματοδοτήσουμε και να αποφασίσουμε ε, τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα έργα. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Ε, δεν αφορά αυτό μόνο τη διαστημική πολιτική, αφορά και αυτά που λέγαμε σε άλλα ζητήματα. Αν δεν λύσουμε ικανοποιητικά το θέμα αυτό, μπορεί να Είμαστε εξαρτημένοι στο τέλος σε τεχνολογίες ε, σημαντικές. Θα εξαρτηθούμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένας δρόμος είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Ο εισηγητής το λέει αυτό το πράγμα. Δεν εννοούμε εδώ μόνο τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, ε, Κίνα, Ινδία και άλλοι. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι στην έκθεσή μας λέμε, το λέει και στον τίτλο, στρατηγική, διαστημική που στην υπηρεσία του πολίτη λέει. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, να ενημερωθούν και οι πολίτες. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ε, να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου που ασχολείται με άλλα προβλήματα τώρα. Αλλά αν, δεν, ε, αν παραιτηθούμε από τα φιλόδοξα σχέδιά μας, αυτό τι επιπτώσεις θα έχει. Τέλος, σου, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και θα, προσπαθήσω να καταθέσω και κάποιες τροπολογίες στο πνεύμα των όσων είπα. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Ταρσνόφσκι. Η κυρία. Όχι, ο κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τους προλαλήσαντες θα είμαι σύντομος, γιατί πολλά ελέγχθησαν ήδη. Συμφωνώ και εγώ με εκείνους που αξιολογούν πολύ θετικά το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι ε, τα λέει τα πιο σημαντικά η έκθεση. Θα ήθελα επίσης ε, να συμφωνήσω με τον κύριο Γκλάντε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα ε, χρηματοδοτικά θέματα. Δύσκολο και περίπλοκο το θέμα, αλλά δεν μπορεί να περιοριζόμαστε μόνο να λέμε ότι μας λείπουν οι πόροι, μας λείπουν οι πιστώσεις για τις ε, θεμελιώδεις λειτουργίες αυτών των έργων. Γιατί όταν κάτι είναι πραγματικά κοινοτικό στα έργα αυτά, ε, αυτό είναι αυτό το μεγάλο έργο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να πραγματοποιηθεί αυτόνομα από κανένα κράτος με, μέλος από μόνο του. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνενώνει τις δυνάμεις για κάτι τέτοιο. Οι οικονομικοί πόροι όμως, οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια και επάρκεια, ούτως ώστε να μην πούμε αργότερα ότι λείπουν πόροι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο με τη σημερινή κρίση να ζητάμε χρήματα από κάποια ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Στο άρθρο 22, στο σημείο 22, γίνεται λόγος για τις εφαρμογές. Η επιτυχία του έργου εξαρτάται από τις εφαρμογές που θα γίνουν στον κύκλο ζωής ε, του έργου. Μπορεί να προσθεθούν πράγματα που δεν τα γνωρίζομαι. Επίσης, ε, θα είναι σημαντικές οι ικανότητες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχία. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει, υπάρχει μια τεράστια υποδομή και η δικιά μας η δουλειά ποια είναι. Να ε, αξιοποιηθούν όλες οι προσφορές στο έπακρο. Εδώ υπάρχει κάτι που το συζητούσαμε ε, πολύ η σύνδεση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ανεξάρτητα από το πώς θα ονομαστεί στο μέλλον το πρόγραμμα αυτό, εμείς θέλουμε επιστημονικές ικανότητες να τις συγκεντρώσουμε, να τις εστιάσουμε εδώ. Υπάρχουν πολλοί τομεί που ακόμα δεν μας έχουν απασχολήσει. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γκλάντε και σχετικά με τη συζήτηση επιμελλοντικών εφαρμογών. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα αυτό, γιατί πρόκειται για τον έλεγχο των δορυφόρων για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και αυτό είναι λογικό να γίνει, γιατί αποτελεί μια μελλοντική προοπτική. Και εγώ θέλω να ε, συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Οι προσπάθειές μας να αναβαθμίσουμε τον Γαλιλαίο είναι σημαντικές διότι έτσι θα έχει καλή ε, προβολή προς τα έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνενώσει με αποτελεσματικό τρόπο και πολλές συνέργειες στις δυνάμεις όλων μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Πατριτσέλο για την καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ωραία. Και τώρα ο συνάδελφος Βεμπέρ. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Πατριτσέλο για την εξαιρετική του δουλειά. Θα ήθελα ωστόσο να ενισχυθούν τα συμπεράσματα της εκθεσής του και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το GMES. Θα προβώ και εγώ λοιπόν στην κατάσταση τροπολογιών. Ξέρουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας, έρχεται στην επόμενη φάση και είναι περιορισμένη οικονομική κίνδυνη σε σχέση με αυτούς που θα μπορούσαν να ληφθούν στην φάση της ανάπτυξης. Τώρα, το κόστος στη φάση αυτή νομίζω ότι μπορεί να είναι υποέλεγχο και να παραμείνει έτσι. Θα μπορούσαμε δηλαδή να βασιστούμε στις εμπειρίες από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως ε, αυτά των μετεωρολογικών δορυφόρων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η παράγραφος 16 να ενισχυθεί και να ζητείτε ε, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από την Κομισιόν το σύνολο της χρηματοδότησης του προγράμματος GMES να ενσωματωθεί στο προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης. Πολλοί συνάδελφοι νομίζω είπαν περίπου τα ίδια, γι' αυτό καλό θα ήταν να ενδυναμώσουμε την παράγραφο 16 από κοινού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως υπενθυμίσατε και εσεί, το GMS e έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ε, παρατήρησης της γη και των ε, περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών εφαρμογών Υπάρχουν κοινοτικέ δαπάνε, κατά την άποψή μου, που πραγματικά είναι πολύ πιο συζητήσιμε από τη συγκεκριμένη. Όπω ε, προτείνει και ο ίδιο ο εισηγητή, ε, σε αυτό το στάδιο να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να έχουμε αποφασιστική διακυβέρνηση και διαχείριση. Θα πρότεινα να εκμεταλλευτούμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από Ευρωπαίου φορεί που έχουν ήδη εργαστεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη ως προς το διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει τα μέσα στη διάθεσή της για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Για να διατηρήσει την αυτονομία της η Ένωση βέβαια θα πρέπει να ευνοηθεί η χρήση ευρωπαϊκών εκτοξευτών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνουν προτάσεις συγκεκριμένες για να έχουμε την κατάλληλη στρατηγική στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε την εξίσωση και την προσαρμογή των πόρων ε, στου στόχους. Έτσι θα έχουμε μια πολύ καλή, όχι μόνο διαστημική ε, πολιτική, αλλά πολιτική ανάπτυξη και βιομηχανική πολιτική. Ένα τελευταίο σημείο το ανέφερε και ο συνάδελφος Γκλάντε. Διεθνή συνεργασία και δίσα θέματα έρευνας με άλλους παράγοντες, φορείς ε, Κίνα, Ρωσία, ΙΠΑ. Άκρος ευκταία αυτή η συνεργασία. Θα πρέπει όμως να πραγματοποιηθεί στη βάση του σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητας. Σήμερα οι θεσμικές αγορές των χωρών αυτών είναι εντελώς ε, κλειστές σε ξένες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και στις ευρωπαϊκές. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να είναι αφελής δεν θα πρέπει να είναι η μόνη διαστημική δύναμη που ανοίγει τις θεσμικές της αγορές στο διεθνή ανταγωνισμό, χωρίς να ζητά κάποιο αντάλλαγμα και χωρίς να έχει ε, την αμοιβαιότητα που θα έπρεπε να υπάρχει. Ευχαριστώ. Λάμπερτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και με συγχωρείτε που άργησα, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει το θέμα, αλλά έχουμε στη χώρα μας ε, μια τραπεζική κρίση που πρέπει να τύχει της αμέριστης προσοχής μου. Λοιπόν, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το διάστημα είναι ένας από τους προφανέστερους τομείς όπου θα πρέπει ε, να ε, κινηθούμε ευρωπαϊκά και όχι εθνικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μακρά διαστημική εμπειρία, δεδομένων όμω των επενδύσεων που απαιτούνται. Γνωρίζουμε επίση ότι μόνο στην ευρωπαϊκή κλίμακα μπορεί κάτι να γίνει. Μόνο αυτή είναι η κατάλληλη κλίμακα. σω να είναι προφανή όλα αυτά, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε και στου πολίτε μα, ότι εδώ πραγματικά η Ευρώπη έχει προστιθέμενη αξία. Δεύτερη παρατήρηση, πιο πολύ θεσμικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε κάποιον εκπρόσωπο τη Κομισιόν εδώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι εντελώς ε, άχρηστο αυτό που κάνει η Επιτροπή μας, διότι μας ε, αφήνουν να μένουμε ε, επιμελώς και σκοπίμως στο σκοτάδι για πολύ σημαντικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη, χρηματοδότηση. Πόσο καιρό ζητάμε σαφή στοιχεία και όχι μόνο κάποιους ε, τίτλους, αλλά θέλουμε στοιχεία αναλυτικά για μικρά προγράμματα όπως είναι το Γαλιλαίο. Μας ε, λένε να παίρνουμε οδηγίες, κατευθύνσεις, συμβουλές ε, σε ό,τι αφορά τη δυστημική πολιτική. Αλλά σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία μας αφήνουν στο σκοτάδι. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι όταν αρχίσαμε να συζητάμε <coughs> τη δημόσια ε, υπηρεσία, ε, τη ρυθμισμένη υπηρεσία του Γκαλιλαίου, α, μας είπε η Κομισιόν, οι περισσότεροι από τους εμπειρονόμες θα είναι στρατιωτικοί. Ενώ είχαν πει αρχικά ότι όχι, είναι μη ε, στρατιωτικού χαρακτήρα έργο, το λέω κατά κύριο Λογάρα, νομίζω ότι στον τομέα αυτό πραγματικά ε, δεν βλέπω να υπάρχει κλίμα συνεργασίας ε, Κομισιών και Κοινοβουλίου, που θα έπρεπε να είμαστε σύμμαχοι μεταξύ μας. Πολλά μένουν κρυφά και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα αποκαλύψουμε. Δεν μιλάμε για πενταροδεκάρες, είναι σημαντικά τα ποσά και θα πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση λογοδοσίας προς, προς τους πολίτες μας ε, για το τι κάνουμε. Αν υπάρχει ένα σχέδιο τώρα που θα έπρεπε να εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Διαστημική και θα πρέπει να το στηρίξουν οι πράσινοι, αυτό δεν είναι άλλο από το GMS. E Γιατί ουσιαστικά καλύπτει μια επιχειρησιακή δυνατότητα που δεν υπάρχει αλλού. Ο Γκαλιλαίο ουσιαστικά πολύ λένε ότι αλληλεπικαλύπτεται με το GPS. Το GMS όμω, Παγκόσμιο Παραγωγή Περιβάλλοντο και Ασφάλεια, είναι κάτι που έχει πραγματικά μια ξεχωριστή προσθέμενη αξία. Και μου φαίνεται λίγο περίεργο η Κομισιόν αποφασίζει να θέσει σε κίνδυνο αυτό το πρόγραμμα. Γιατί α τα πούμε με το όνομά του τα πράγματα. Ο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα η Κομισιόν ουσιαστικά τι κάνει, ε, οθεί στην ε, εξαφάνιση, στην εξάλληψη το GMS και οθεί, προωθεί άλλα πράγματα το, ε, Γαλιλαίο για παράδειγμα, ή και το ίτερ. Προσπαθεί να τα κρατήσει στη ζωή. Το GMS e οικονομικό, είναι προβλέψιμο, είναι ασφαλέ, θα έλεγα και αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το πει κανεί για το ίτερ. Και δεν θα περίμενα να έρθει η Κομισιόν εδώ να μα πει ότι ε, το ίτερ είναι στο διάστημα και δεν ξέρουμε να το κάνουμε γιατί το αφήνουμε λοιπόν εκτό του προπολογισμού, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εντό του προπολογισμού και κρατάμε το GMS e και το Galileo έστω και αν είναι κάπως ε, περιοριστική η όρη του. Αλλά τελικά τι θέλει να πει η Κομισιόν ε, αφήνοντας εκτός το GMS, ότι μάλλον δεν το θέλει. Αυτό είναι τρελό. Ένα σχέδιο που γεννά αξία, όπου μπορούμε να εντοπίσουμε ξεκάθαρα ε, ποιες επενδύσεις απαιτούνται για το GMS. Αυτό λοιπόν το πετάμε έξω και για άλλα προγράμματα που δεν ξέρουμε, σίγουρα σύντομα δεν θα έχει κάποια προσθέμενη αξία και μιλάω για το ITER, που έχει ένα ε, ε, κόστος εντελώς εκτός ελέγχου και απρόβλεπτο το κρατάμε. Ποιος μάνατζερ θα μπορούσε να πλασάρει κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενό τέτοιου μάνατζερ, γιατί πάνω από 30 δευτερόλεπτα δεν θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτού. Το κάνει όμω η Κομισιόν και το κάνουν τα κρατημέλη. Λε και δεν λογοδοτούν στου πολίτε του. Και στη χώρα μας έχουμε ε, να εξοικονομήσουμε δέκα δις ε, λόγω περικοπών ε, στις δημόσιες δαπάνες του χρόνου. Θέλω και τα άλλα κράτη-μέλη να πάνε στα κράτη-μέλη και να πούνε ότι θέλουμε να χαλάσουμε για το Ίτερ και για τον Καλλιλέο πάρα πολλά πόσα, χωρίς όμως να έχουμε κάποιο καθορισμένο αποτέλεσμα προεξοφλημένο. Λοιπόν, εμένω στη θέση μου, αν δεν έχουμε σαφή ε, στοιχεία και θέλω κόστος, ανάλυση κόστους ωφέλους για το ίτερ, Θέλω να δω ποιο είναι το κόστος, ποια είναι τα ωφέλη. Δεν έχει για μας κανένα όφελος το ίτερ. Θα πρέπει να δούμε τώρα το Γαλιλαίο, το πρόγραμμα αυτό. Τι ωφέλη μπορεί να προσφέρει απέναντι στο κόστος. Μέχρι στιγμής μας έχει αφήσει στο σκοτάδι κομισιόν. Δεν μας έχουν ενημερώσει επισήμως καθόλου για τον Γαλιλαίο. Τώρα, επιτυχέ έρευνα και ανάπτυξη διαστημική πολιτική. Εμεί το έχουμε πει ξεκάθαρο. Όταν περάσουμε στη βιομηχανική φάση, δεν θα πρέπει να ε, φύγουν χρήματα από το προπολογισμό τη ε, έρευνα και τη καινοτομία, γιατί πλέον μιλάμε για τη βιομηχανική πολιτική. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πτυχέ έρευνα και καινοτομία στον Καλλιλέο ή στο GMES. Φυσικά και πρέπει να, δια, ε, να χρηματοδοτηθεί η διαστηριότητα από τον προπολογισμό ε, του, 2020. Απλά θέλω οι διαστημικές πτυχές να ληφθούν υπόψη όπως και οι τεχνολογίες των πληροφοριών ως μια τεχνολογία που επιτρέπει ε, χρήσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, που μας διευκολύνει να αντιμετωπίσουμε κάποιες κοινωνικές αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει η διαστημική ε, συνιστόσα. Μπορεί το GMS να μας βοηθήσει να μεταρρυθμίσουμε και την γεωργική μας πολιτική, για παράδειγμα. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Και έρχομαι σε μια τελευταία παρατήρηση ό,τι αφορά τη στρατιωτική πτυχή. Δεν είμαι αφελή, θα τα πω ξεκάθαρα. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ενόπλε δυνάμει και ξέρουμε ότι και το διάστημα είναι ένα εργαλείο που ίσω χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί από τι ε, στρατιωτικέ δυνάμει ε, για στόχου συλλογής πληροφοριών, επικοινωνίας, επιτήρησης, ε, εποπτεία κτλ. Τι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει οι στρατιωτικέ πτυχέ του Γκαλιλαίο ή ακόμη δυνητικό και του GMS να χρηματοδοτηθούν από προπολογισμό εκτό του αμυντικού προπολογισμού. Δηλαδή, με άλλα λόγια. Βρείτε μου επιχειρήματα ε, που δείχνουν ότι έχουμε στατιωτικά ωφέλη. Αλλά ότι το μερίδιο του προπολογισμού πρέπει να προέρχεται από τους προπολογισμούς τους αμυντικούς των κρατών μελών. Αν θέλουν ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Άμυνα, κανένα πρόβλημα. Αλλά πάλι θα πρέπει οι προπολογισμοί να προέρχονται από μέλη και να ρέουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να αλωνίζουν οι στρατιωτικές δυνάμεις με την ε, διαστημική πολιτική. Δεν λέω ότι πρέπει να βάλουμε βέτο στη στρατιωτική χρήση, αλλά αυτός που χρησιμοποιεί πρέπει και να πληρώνει. Αυτή είναι η βασική αρχή την οποία πρέπει νομίζω να στηρίξουμε. Ρωτώ την Κομισιόν, τον κύριο Γκονζάλες, θέλει να μιλήσει για την Κομισιόν, κύριε Γκονζάλες ή κάποιος άλλος υπεύθυνο. Ευχαριστώ. Σημειώσαμε ότι η έκθεση υποστηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, και επίσης ε, σημειώσαμε και τα διάφορα σχόλια που έγιναν ε, και μάλιστα κυρίως όσα αφορούν τη χρηματοδότηση του GMS. Δεν νομίζω ότι θα επανέλθω σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο γιατί η Κομισιόν ήδη έχει τοποθετηθεί σχετικά. Και γιατί αποφάσισε να προτείνει να χρηματοθετηθεί εκτός ε, του προβλήματος τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Θέλω όμως να επανέλθω στο σχόλιο σχετικά με την ε, έλλειψη διαφάνεια και ε, με την έλλειψη αριθμητικών στοιχείων. Να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν κατέθεσε την έκθεσή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων ε, δορυφορικής μεδιπλοήγησης φέτος τον Ιανουάριο και αναφέρεται συγκεκριμένα και στο Γαλιλαίο. Φυσικά η ανακοίνωση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ξορισμού ε, περιλαμβάνει μεγάλους τομείς του προπολογισμού. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά η πρόταση για σχέδιο κανονισμού θα κατατεθεί σύντομα από την Κομισιόν και για το Γαλιλαίο και για το GMS. E αυτοί οι κανονισμοί, τα σχέδια κανονισμών θα συνοδεύονται και από μελέτες αντικτύπου που θα αναφέρουν λεπτομερώς το business case και για τα δύο προγράμματα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου θα δουν ότι δεν ε, υπάρχει απόπειρα απόκρυψης ε, της οικονομικής ε, λογικής που διέπει τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να καταστήσω σαφή τη θέση της Κομισιόν. Είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε να ανταλλάσσουμε αριθμητικά στοιχεία και διαθέσιμες πληροφορίες και να αιτιολογούμε με τον κατάλληλο τρόπο το κόστος των προγραμμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πατρετσέλο θέλει να προσθέσει κάτι, ορίστε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδελφούς ε, για τις ε, παρεμβάσεις τους. Φυσικά αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να βελτιωθεί με την κατάσταση και με όλες ε, τις σκέψεις που θα κάνουμε από κοινού. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ σε μια σημαντική πτυχή που αναφέρθηκε ε, σχετικά με την αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Πρόκειται για ένα στοιχείο σημαντικό για μας, γιατί μια αυτόνομη διαστημική πολιτική δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και μια στρατηγική με πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς φορείς. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια τεχνολογία και μια αυτονομία σε ό,τι αφορά και τους δορυφόρους. Γιατί αποτελούν ε, ενσωματωμένο τμήμα της όλης στρατηγικής Τώρα υπήρξε και το θέμα της χρηματοδότησης που αναφερθήκε από τους συναδέλφους και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο, είναι το πιο σημαντικό. Η Κομισιόν ε, είπε ότι έχει τοποθετηθεί ήδη για, ε, για το θέμα της ε, χρηματοδότησης του GMS. E Όμως εμείς ως Επιτροπή ήτρε πρέπει να κάνουμε και τη δική μας αξιολόγηση και να αναπτύξουμε το δικό μας προβληματισμό σχετικά με το θέμα αυτό. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε τις επόμενες εβδομάδες να καταλήξουμε σε ένα κείμενο συμπεφωνημένο και το οποίο θα μπορεί να προσδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία όθηση για την ε, πολιτική διαστήματος που είναι στρατηγική σημασία και για την Ένωση και για τις διάφορες χώρες και κυρίως για το βιομηχανικό κόσμο. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα σε αυτή την στιγμή κρίση, σε αυτούς τους καιρούς της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στα διάφορα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν μία νέα όθηση αυτού του τομέα θα μπορούσε ε, να βοηθήσει και την ανάπτυξη της οικονομίας. Και μάλιστα μπορεί να δημιουργηθούν και νέες θέσει εργασία με το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να δοθεί νέα όθηση. 30 δευτερόλεπτα στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Η έκθεση που δημοσίευσετε νωρίτερα αυτό το έτος ήταν άδεια. Εσείς είπατε ήταν γεμάτη αριθμητικά στοιχεία. Εγώ όμως αυτά τα στοιχεία τα είδα επίσημα. Έτσι λοιπόν θα λάβετε γραπτό ερώτημα από μένα σήμερα το απόγευμα. Θέλω τη δέσμευσή σας ότι θα αποκαλύψετε πλήρως, θα δημόσετε πλήρως πώς καταλήξατε ε, στο ένα δισεκατομμύριο το χρόνο, πώς καταλήξατε σε αυτή την εκτίμηση. Και αν εσείς είστε έτοιμος να το πράξετε αυτό, πολύ ωραία. Äh, Εντάξει. Θα περιμένουμε την ερώτηση και τις απαντήσεις. 12 Οκτωβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Μετά θα γίνει η δεύτερη διαβούλευση. Ευχαριστώ. Κλείνουμε την ημερήσια διάταξη και το απόγευμα θα έχουμε ένα εξαιρετικό hearing στο οποίο είστε όλοι προσκεκλημένοι.